Καλησπέρα σας κύριε και, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Και πριν περάσουμε στο κυρίως θέμα της απογευματινής μας συνεδρίασης, την ανταλλαγή δηλαδή απόψεων με τον Αμερικανό Υπουργό Γεωργίας, πριν λοιπόν να περάσω στο καλωσόρισμα προς τον Υπουργό, να δούμε κάποια διαδικαστικά. Καταρχήν να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Το σημείο 13 θα συζητηθεί... Yeah. Συγγνώμη που σε διακόπτω κύριε Πρόεδρε, λέει χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Δεν ακούμε τη διερμηνία από τα αγγλικά. Now is okay. Okay. We can start. Εντάξει τώρα. Επαναλαμβάνω, θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Το σημείο 13 θα το συζητήσουμε μετά το 6. Σε ό,τι αφορά το σημείο 7, δηλαδή την ψηφοφορία για τα έκτακτα εμπορικά μέτρα για την Τινησία, πάλι έχουμε πρόβλημα τεχνικό. Now, I think that now okay. Okay. Επαναλαμβάνω, το σημείο 13 θα το συζητήσουμε πριν το 16 και το σημείο 7, την ψηφοφορία, την αναβάλουμε για τη συνεδρίαση της 11 Ιανουαρίου. Σήμερα θα εξετάσουμε μόνο τις τροπολογίες. Έχουμε και απευθεία αναμετάδοση τη συνεδρίασή μα. Διερμηνία υπάρχει σε 20 γλώσσε με εξαίρεση εστονικά, μαλτέζικα, σλοβακικά και κελτικά και σα ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Επίση, να σα υπενθυμίσω ότι την επόμενη Πέμπτη μεταξύ 9.30 και 10.30 θα έχουμε την έκτακτη συνεδρία τη Επιτροπή Γεωργία με θέμα ανταλλαγή απόψεων με τον ειδικό ε, πρέσβη της ΦΑΟ επευκαιρία του Διεθνούς Έτους ε, του Εδάφους και μάλιστα θα έχουμε κοινή συνεδρίαση των τριών επιτροπών Γεωργίας, Περιβάλλοντος και ανάπτυξη για την ανταλλαγή απόψε με τον ειδικό πρέσβη της ΦΑΟ. Επίσης να σας προσκαλέσω σε μια έκθεση επευκαιρία του Διεθνού Έτους για το εδάφη που οργανώνει η ΦΑΟ στον τρίτο όροφο του κτηρίου Αλθιέρο Σπινέλη που βρίσκεται απέναντι. Αυτές είναι οι κυριότερες ανακοινώσεις που είχα να κάνω. Μην ξεχνάτε και το σεμινάριο που οργανώνουμε στις 9 Δεκεμβρίου, αλλά έχουμε γι' αυτό χρόνο. Περνάμε στο σημείο 3, την έγκριση των πρακτικών, όσοι είστε. Και μετά από αυτές τις τεχνικές ανακοινώσεις, θα ήθελα να περάσουμε στο κυρίω θέμα, που όπως σας είπα είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Αμερικανό Υπουργό Γεωργίας, τον οποίο έχω την τιμή να καλωσορίζω στη συνεδρίασή μας. Τον ευχαριστώ θερμά που δέχτηκε την πρόσκληση της Επιτροπής Γεωργίας, προκειμένου να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για θέματα γεωργίας. Η παρουσία σας μας δίνει και μια ιδανική ευκαιρία για να ανταλλάξουμε μεταξύ μας απόψεις και να ενημερωθούμε απευθείας από πρώτο χέρι από σας Θεωρώ ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων στην ε, κρίσιμη αυτή στιγμή είναι πολύ σημαντική, γιατί ε, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι γίνονται πολύ σοβαρές συζητήσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, τη TIP. Γι' αυτό και είναι πολύ επίκαιρη αυτή η ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε μια σύγκληση. Γνωρίζουμε ότι είστε πολύπειρος ε, σε θέματα γεωρικής πολιτικής και είστε στενός συνεργάτης του Προέδρου Ομπάμα και μάλιστα αναλάβατε το Υπουργείο Γεωργίας από την αρχή της Προεδρικής Αιτίας του κ. Ομπάμα. Έχετε πολύχρονη και πλούσια πείρα λοιπόν στα θέματα της γεωργίας και γι' αυτό περιμένουμε την δική σας ε, παρουσίαση που γίνεται υπό τη σκοπιά μιας μακροχρόνιας και πλούσιας πείρας, όπως σας είπα, για τα γεωργικά ζητήματα. Αφού ακούσουμε τη δική σας ομιλία, θα έχουμε και μια ανταλλαγή απόψεων με τους ευρωβουλευτές και έτσι θα επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά θέματα για μας, ε, επευκαιρία της διατλαντικής σχέσης ε, εμπορίου και επενδύσεων και θα εξετάσουμε και τις σημαντικές αναπτυξιακές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ίσως αυτή η συμφωνία του TTIP θα αποτελέσει το πρότυπο για εμπορικές συμφωνίες ε, σε θέματα δασμολογικά, σε θέματα τελωνιακά, σε θέματα υγειονομικά και μπορεί να γίνει πρότυπο τέτοιων εμπορικών συμφωνιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ, σας καλωσορίζω και πάλι στη συνεδρίαση και σας δίνω το λόγο. Uh, uh, uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια που ακούσαμε στην εισαγωγή σας. Εκτιμώ πολύ την δυνατότητα που μου δίνεται μέσω της προσκλήσεως μιλήσω. Ευχαριστώ τα μέλη που ήρθαν εδώ σήμερα που μου δίνετε το χρόνο σας και τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως ερχόμουν από το αεροδρόμιο σήμερα το πρωί, δεν μπορούσα να σκεφτώ μία από τις πρώτες μου επισκέψεις στην Ευρώπη. Τότε ήμουν κυβερνήτης της πολιτείας της Άιουα ταξίδεψα στη Γαλλία με τον κυβερνήτη της Οκλαχώμα και τις γυναίκες μας και σκοπός της επίσκεψης ήταν να θεωρήσουμε τις υποχρεώσεις που είχαν λάβει οι Γάλλοι προς τους ε, νέους τους. Ε, Ήθαμε να κάνουμε το ίδιο και εμείς. Αναγνωρίσαμε τη σημασία που έχουν τα νέα παιδιά, η παιδεία των παιδιών. Ήταν ε, συνεδρίαση αρχή το πρωί, ήταν ώρα για, να, για ένα, πάρουμε ένα μεζέ και ο κυβερνήτης του Κλαχώμα και εγώ εκπλαγήκαμε όταν ε, δώσανε φρούτα και λαχανικά όταν ήρθαν οι Κινέζοι ε, σε παιδιά 3-4 ετών. Και η γυναίκα μου και εγώ δεν θα είχαμε αναθέσει ε, τα παιδιά μας 3-4 ετών στην Κίνα στους Κινέζους και είχαμε όμως χαρεί πάρα πολύ με την ποιότητα των παιδιών. Και μου είπαν ότι πόσο μεγάλος ο βρασμός. Και τους, δίσα, τους δώσανε λοιπόν τα φαγητά αυτά σε σερβίτσιο πορσελάνινο. Και τώρα προσπαθούμε για μία ακόμη φορά να επαναλάβουμε αυτή την προσπάθεια με την πρωτοβουλία για τα νέα και υγιή παιδιά και η Μισελ Ομπάμα, η γυναίκα του Προέδρου, ανέλαβε και πρόθεσε το θέμα. Θέλουμε οι νέοι μα να τρέφονται καλά και να έχουν μια καλή αρχή στη ζωή του. Με εντυπωσιάζει λοιπόν το γεγονό ότι πολύ συχνά ε, μοιάζουμε από ό,τι διαφέρουμε όσον αφορά τα θέματα γεωργία και τροφίμων και χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψει ούτω ώστε να υπογραμμίσουμε περαιτέρω αυτή την αρχή. Να πω λοιπόν ότι πράγματι και κυρίως οι γεωργοί της χώρα μου Είμαστε, μοιάζουμε πολύ με τους γεωργούς της Ευρώπης, με τους γεωργούς. Οι γεωργοί και εδώ και στην ΣΥΠΑ είναι περήφανοι για τις ρίζες τους, πιστεύουν στη σκληρή δουλειά, πιστεύουν στην ε, βιωσιμότητα, καταλαβαίνουν την ευθύνα και το καθήκον που έχουν απέναντι στις μελλοντικέ γενιές για να, ε, να οργώσουν τη γη και να παράγουν τρόφιμα είναι υπερήφανοι διότι μπορούν να θρέψουν όχι μόνο το λαό της χώρας τους αλλά σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζουν ότι έχουν μια ευθύνη όσον αφορά την ε, ασφάλεια των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο όπως κάθε γεωργός σε κάθε χώρα ενδιαφέρονται για νέες δυνατότητες σε αναπτυσσόμενες αγορές αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα παραγωγής τροφίμων με την αλλαγή του κλίματος θα γίνει όλο και πιο δύσκολο. Το θέμα της αλλαγής του κλίματος είναι κάτι που θα συζητήσουμε σε δύο μέρες στο Παρίσι όταν θα μεταβώ εκεί για να συμμετάσχω στις εργασίες του COP21 και θα παρουσιάσω τα βήματα που κάνουμε στις ΗΠΑ στη Γεωργία για να μειώσουμε τις εκπομπές μας και να έχουμε παραγωγή βιώσιμη και νομίζω ότι μπορούμε να διπλασιάσουμε τη μείωση των εκπομπών στη Γεωργία επιθελοντικής ε, βάσεως. Οι γεωργοί μας, όπως ισχύει και στην Ευρώπη, νομίζω ότι αντιμετωπίζουν την αλλαγή του κλίματος. Επίσης έχουν προβλήματα με την αλλαγή του γούστου των καταναλωτών και την ανάγκη που υπάρχει για νέα προϊόντα και γι' αυτό η γεωργία απαιτεί μια ευελιξία και καινοτομία. Ένα μήνυμα που θα ήθελα να παρουσιάσω στην ομάδα σήμερα είναι ότι η Αμερικανική γεωργία πολύ συχνά δεν γίνεται καλά αντιληπτή στις ΗΠΑ και ίσως δεν είναι και τόσο ευληπτικές στο εξωτερικό Κάποιοι στη ΣΥΠΑ πιστεύουν ότι η Αμερικανική Γεωργία είναι μια μεγάλη επιχείρηση παραγωγής ενία. Δεν ισχύει αυτό. Κατάγουν μια πολιτεία που έχει συνήθως οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και μικρές εκμεταλλεύσεις. Εμείς στο Υπουργείο Γεωργίας, τα τελευταία χρόνια που ήμουν Υπουργός Γεωργίας της ΕΠΑ, εστιαστήκαμε κυρίως στην ενθάρρυνση μεγαλύτερης ποικιλομορφίας στην Αμερικανική Γεωργία αληθεύει ότι πολλοί γεωργοί στη ΣΥΠΑ χρησιμοποιούν γενετικά τροπημένες καλλιέργειες, αλλά επίσης αληθεύει ότι άλλοι γεωργοί και αυξανόμενος αριθμός αυτών ε, παράγουν βιολογικά προϊόντα και χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακές μεθόδους ε, παραγωγής. Σίγουρα αληθεύει ότι έχουμε ποικιλομορφία στα προϊόντα που παράγουμε, από εξειδικευμένα προϊόντα μέχρι τι παραδοσιακές καλλιέργειες και ε, προσπαθούμε να συντηρήσουμε και κάποια προϊόντα. Υπάρχει ποικιλία των εκμεταλλεύσεων σε μέγεθος. Έχουμε, τα βάλουμε επιθετικές προσπάθειες να ενθαρρύνουμε την τοπική παραγωγή στη ΣΥΠΑ ε, με 5, 15, 60 στρέμματα περίπου και προσπαθούμε να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να μπουν στην ε, γεωργία στην Αμερική. Ελπίζω κατά τη διάρκεια λοιπόν τη σημερινή επισκέψεω να ενθαρρύνω την εξή έννοια, δηλαδή ότι η Αμερικανική Γεωργία δεν είναι μονολυθική, αλλά έχει μεγάλη ποικιλομορφία σαν παραγωγή. Όλοι αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του κόσμου σε τρόφιμα και αυξάνεται ο πληθυσμό στον κόσμο. Εκτιμάται ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή ε, κατά 60-70 χρόνια, ε, κατά 60-70% σε 30-40 χρόνια και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα δε περισσότερο είναι προβληματικό με την αλλαγή του κλίματος. Γι' αυτό η άρχισαν να βλέπουν τρόπους με τους οποίους μέσω έρευνας μπορούμε να δημιουργήσουμε καινοτομίε που θα μας επιτρέψουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα και γι' αυτό αστερνθήκαμε ακριβή γεωργία αναγνωρίζοντας ότι κάθε στρέμα γης που καλλιεργείται δεν είναι το ίδιο με γειτονικό ε, κτήμα, γειτονική έκταση και βλέπουμε ποια είναι, ποιος είναι ο χαρακτήρας κάθε έκτασης και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τι σπόρους να χρησιμοποιήσουμε, πόσα λιπάσματα χρησιμοποιήσουμε, τι χημικά να βάλουμε, αν βάλουμε χημικά ε, και πώς να προστατεύσουμε τις σπάνιες πηγές ύδατος μέσω ακριβής, ακριβούς καλλιέργειας αναγνωρίζουμε ότι το θέμα δεν είναι να αυξήσουμε την παραγωγή, αλλά να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα τρόφιμα που χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό μαζί με πολλές άλλες χώρες ζητούμε και εμείς διεθνείς προσπάθειες για την μείωση ε, της πατάλης ε, τροφίμων. Σχεδόν ένα τρίτο από τα τρόφιμα παράγοντες παταλώνται για ποικίλου λόγους. Τη είπα πολύ συχνά, διότι έχουμε πάρα πολλά, τρώμε πολύ, και δεν μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε ή να ανακυκλώσουμε τα τρόφιμα σε αναπτυσσόμενε χώρε, ίσω ε, να μην είναι σωστή αποθήκευση και γίνεται σπατάλη τροφίμων. Τέλο πάντων, υπάρχει παγκόσμια ανάγκη να εστιαστούμε επί ε, μειώσεω τη σπατάλη των τροφίμων και πιστεύουμε ότι ένα κομμάτι τη ασφαλεία τη επισητιστική καλύπτεται μέσω και συμφωνιών για δίκαιο εμπόριο. Στη ΣΥΠΑ θεωρούμε ότι οι εμπορικέ συμφωνίε παρέχουν μια σταθεροποίηση όσον αφορά τι τιμέ των ε, προϊόντων και για το εισόδημα των γεωργών. Δημιουργούνται θέσει απασχόληση. Πάνω από ένα εκατομμύριο δουλειέ σχετίζονται άμεσα με τι εξαγωγέ γεωργιών ε, από τα 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια θέσει απασχόληση σχετίζονται με τι εξαγωγέ. Προωθείται η καινοτομία και ενισχύει και τι σχέσει. Είχαμε κάποιε εμπειρίε με αυτό ε, την ε, Συμφωνία Ελευθερου για τη Βόρεια Αμερική με την έκπληξη ε, είδα πώς είχαν κάνει τις χώρες τη Συμφωνία στη Γεωργία, το Μεξικό, Καναδάς και Ηνωμένε Πολιτείε, όλες είδαν αύξηση στις εμπορικές συναλλαγές και ήταν ε, ισορροπημένε οι σχέσεις. Είχαν ευκαιρίες οι Γεωργοί να ωφεληθούν και στις χώρες. Πρόσφατα συνήψαμε ε, τις ολοκληρώσουμε διαπραγματεύσεις για την ε, συμφωνία του ειρηνικού, την εμπορική, δημιουργεί δυνατότητε όχι μόνο για τα μέλη του TPP αυτής της συμφωνία και για τους Αμερικανούς, αλλά και για τους γεωργού στην Ευρώπη να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες με τις μέσει τάξεις Αυξάνεται πολύ η μεσαία τάξη στην Κίνα, περίπου 535 εκατομμύρια καταναλωτέ είναι στη μεσαία τάξη στην Ασία σε 15 χρόνια. Μπορεί να αυξηθεί κατά 2,7 δισεκατομμύρια ανθρώπου σε αυτή η τάξη, δημιουργηθούν πολλέ ευκαιρίε για τους σε όλο τον κόσμο. Και πιστεύουμε ότι οι διαπραγματεύσει για αυτή τη συμφωνία του ειρηνικού δημιουργεί τη δυνατότητα να δώσουμε όθηση στις συνομιλίε που θα διεξαχθούν και με τους Ευρωπαίους ε, στα πλαίσια του TTIP, στι διαπραγματεύσει του TTIP. Ε, πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά φέλη και για, την, ε, για τη ΣΥΠΑ και για την Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και σοβαρές προκλήσεις και προβλήματα. Κάποιες δυσκολότατες ε, αποφάσεις που να ληφθούν μετά από δυσχερέστατες συνομιλίες. Προσεγγίζουμε την ασφάλεια των τροφίμων με κάπως διαφορετικό τρόπο. Γίνονται συζητήσεις εδώ για την αρχή της προλήψεως της ΣΥΠΑ. Είναι μια αξιολόγηση που γίνεται μέσα στον κίνδυνο. Πολύ συχνά αυτά θεωρούνται ότι είναι διαφορετικά, αλλά στην πράξη όλα αυτά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή ασφαλή τρόφιμα για κατανάλωση. Κατανοούμε ότι υπάρχει μια ανάγκη για προστασία, για προτάσεις που δίνουν προστιθέμενη αξία. Πολύ συχνά αυτό αφορά το πού καλλιεργείται ένα προϊόν, ε, σε ποια γεωγραφική περιοχή, Όλοι θα έχετε γεωγραφικές ενδείξεις που δίνουν μια προστασία προς τη της αξίας. Εμείς έχουμε εμπορικά σήματα στη ΣΥΠΑ. Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα, αλλά ο στόχος είναι ο ίδιος. Θέλουμε να παράσχουμε ε, προστασία για να έχουμε τη θέμενη αξία. Να γνωρίζουμε ότι στον τομέα των κανονισμών για, τα, για την υγειονομία και τα φυτογειονομικά η επιστήμη πρέπει να θέτει προδιαγραφές επιστημονικές για να επικρατεί προβλεψιμότητα και διαφάνεια σε πολλές χώρες. Πρόσφατα επέστρεψα από την Κίνα όπου γίνεται συζητήση για ευρύ φάσμα ανησυχιών ε, που αφορούν τους διάφορους κανονισμούς για τα υγειονομικά, φυτονομικά και διάφορες πολιτικές πτυχές. Ε, όλα αυτά ε, δημιουργούν δυσκολίες για μας. Προφανώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των συστημάτων μας, αλλά το βασικό μήνυμα που θα ήθελα να σας μεταδώσω είναι ότι κατά την άποψή μου δεν αφορά το να έχουμε ταυτόσιμα συστήματα αλλά ισοδύναμα και μπορούμε να πετύχουμε τον ίδιο στόχο χρησιμοποιώντας διαφορετικές ρίζες και διαδρόμους από τη στιγμή που έχουμε κοινό στόχο και νομίζω ότι ο στόχος είναι ίδιος να έχουμε επαρκή εφοδιασμό τροφίμων που παράγεται με βιώσιμο τρόπο το τρόφιμο, να είναι ασφαλές προς κατανάλωση και να καλύπτονται οι ανάγκες των λαών μας και να καλύψουμε τις αυξανόμενες ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού του κόσμου Προφανώς εκτιμούμε τα ευρωπαϊκά προέντα στη ΣΥΠΑ, ας πούμε κρασί και τυριά πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ ε, τυριού και ε, κρασί από την Ευρώπη καταναλώνονται στην ε, Αμερική και αν εφαρμοστεί το TTIP πιστεύω ότι σίγουρα δεν θα μειωθεί αυτός ο αριθμός και πιθανότατα θα αυξηθεί αυτό αντίθεται με τα 500 εκατομμύρια ευρώ των ε, ε, αμερικανικών τυριών και κρασιών που πολλούνται στην Ευρώπη. Υπάρχει εδώ δυνατότητα για συνεχιζόμενη, για, αύξηση των πωλήσεων των ευρωπαϊκών προϊόντων στη ΣΥΠΑ και να δημιουργηθούν δυνατότητες και ΗΠΑ να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν σε αυτή την αγορά, αλλά στο τέλος οι καταναλωτές τελικά θα κάνουν τη σωστή επιλογή από μόνοι τους και ελπίζω πραγματικά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον να τους δώσουμε την επιλογή είναι ενδιαφέρουσε οι συζητήσει και σίγουρα θα ακουστούν κάποια σχόλια και ερωτήσει για διάφορα θέματα που θα έχετε. Θα ήθελα να κλεισω λέγοντα λέγοντας ένα-δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα η Αμερικανική Γεωργία πραγματικά είναι ποικιλόμορφη, ε, πράγματι δεν είναι μόνο λυθική και σε πολλέ περιπτώσει εξελίσσεται και μεταλλάσσεται ένα σύστημα που παρέχει δυνατότητες για μεγάλη παραγωγή, παραγωγή μεγάλης κλίμακας αλλά και για μικρές εκμεταλλεύσεις. Έχουμε αμοιβέ ευθύνε όσον αφορά την ασφάλεια τροφίμων στον κόσμο. Πρέπει να καλυφθούν εν μέρη μέσω επιστήμη, εν μέρη μέσω ακριβού γεωργία και εν μέρη μέσω αποφυγή τη πατάλη. Αλλά οι εμπορικέ αυτέ συμφωνίε έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν. Και τέλο, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μας ε, δεν αυταπατώμε, ξέρω ότι θα είναι δυσχερέστατε. Ελπίζω όμω ότι θέλουμε πράγματι να βρούμε έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα απαιτούμε ένας από τον άλλον να έχουμε ταυτόσημα ίδια συστήματα, αλλά αντίστοιχα συστήματα ισοδύναμου που τελικά πετυχαίνουν τον ίδιο στόχο με διαφορετικό τρόπο και μέσω διαφορετικής διαδρομής. Οι καταναλωτές μας θα ωφεληθούν και οι θέσει απασχόληση θα ωφεληθούν, οι γεωργοί μα θα ωφεληθούν και οι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Ηνωμένων θα ενισχυθούν. Και όπω πρότεινε και ο Πρόεδρο, και θα κλείσω εδώ, όπω πρότεινε ο Πρόεδρο, δεν είναι αυτό μια συμφωνία που αφορά μόνο τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά υψηλέ προδιαγραφέ, αφορά την αποστολή μηνύματο προ τον υπόλοιπο κόσμο σχετικά με την εμπορική συμφωνία υψηλή ποιότητα, τι μορφή πρέπει να έχει, τι πρέπει να περιέχει. Δεν γίνεται ένα αγώνα προ τον ε, ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Πρέπει να ηγηθούμε να δώσουμε το παράδειγμα στον υπόλοιπο κόσμο και προσβλέπω στα σχόλια των ε, μιλητών σήμερα και να μπορέσω να απαντήσω όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις ε, χρόνο επιτρέποντος. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ως ήθιστε, θα ακούσουμε τώρα τους συντονιστές μας πρώτα, σε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων. Μετά θα απαντήσετε στις ερωτήσεις των συντονιστών και κατόπιν θα έχουμε και ένα δεύτερο γύρο έρωτα απαντήσεων. Δύο λεπτά έχουν οι συντονιστές και ένα λεπτό οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Δυστυχώς ε, δεν μας επιτρέπει παραπάνω ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρώτο ο κύριος ε, Ντες από το ΕΛΚ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας εδώ κύριε Υπουργέ. Εξηγήσατε τα της Αμερικανικής Γεωργίας και είστε διατριμμένος να απαντήσετε σε ερωτήσεις μας. Στα ταξίδια που έχω κάνει στις ΗΠΑ διαπίστωσα ότι ασφαλώς και υπάρχουν μικρές και μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Είδα γεωργική εκμετάλλευση κτηνοτροφική στις ΗΠΑ με 10 αγελάδες. Όμως, κατά μέσον όρο είναι δεκαπλάσιο το μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης στην ε, Αμερική από ότι σε εμά. Δηλαδή είναι τη τάξη των 180 εκταρίων, κατά μέσον όρο. Μεγάλη διαφορά λοιπόν. Διάβασα σε ανακοινωθέν τύπου ότι ψηφίζεται νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα τρισεκατομμύριο περίπου, 965 δισεκατομμύρια δηλαδή, που θα δοθούν τα επόμενα πέντε χρόνια στην ε, Αμερικανική Γεωργία. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι με ποιον τρόπο θα δαπανηθούν τα χρήματα αυτά. Δεν πρόκειται για άμεσε ενισχύσει. Όμω, αν υπολογίσω αναεκτάριο, εκτάριο, πάλι μου βγαίνουν εκεί 400 ευρώ αναεκτάριο. εκτάριο. Άρα βρισκόμαστε και εδώ ε, στα ίσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την TTIP τώρα, την συμφωνία TTIP. Εγώ είμαι υπέρ ε, συμφωνίας με τους Αμερικανούς, όμως υπό τους σωστούς όρους. Ανησυχώ όταν ακούω από τους διαπραγματευτές ότι εξακολουθεί να συζητείται ένα σύστημα αδειών εισαγωγών. Εάν μπει σε εμπορική συμφωνία τέτοιο σύστημα, εγώ δεν θα μπορέσω να διεξηγήσω ποτέ αυτό στους αγρότες μου εδώ και δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούν την συμφωνία αυτή. Μπορώ να δεχτώ κάποια ανώτατα όρια ανώτατα όρια για τις εισαγωγές κάποιων προϊόντων, όχι όμως άδειε για εισαγωγές. Υπάρχει και άλλο θέμα, υπάρχει η σφραγίδα του βιολογικού προϊόντος. Αλλά δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο, ο χρόνος όπως ξέρετε είναι περιορισμένος. Ελπίζω να μου απαντήσετε στις ερωτήσεις που έθεσα. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Δεκάστρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό, τον Τόμ Βίλτσακ που είναι εδώ και παρίσταται για πρώτη φορά. Από ό,τι θυμάμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει το θεσμικό μας όργανο και ήταν χαρά που άκουσα την ομιλία του που έθεσε τόσες στοιχεία όσον αφορά τη Γεωργία στις ΗΠΑ που πολύ συχνά δεν ακούγονται αυτά σε αυτή την αίθουσα, για να υπόψη. Θα προσπαθήσω συντομότατη αυτή η παρέμβαση να θέσω δύο ερωτήσεις. Πρώτη, που αφορά τη Διατλαντική αυτή συμφωνία αυτή η Επιτροπή με τον συνάδελφο Jim Nicholson ετοίμασε γνωμοδότηση και ψηφίσαμε γνωμοδότηση που θέτει κάποιες ε, σκέψεις όσον αφορά τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που η Διατλαντική συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει τους Γεωργούς. Ένα σημείο θέλω να θίξω μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουμε το 1 τρίτο των διεθνών, των παγκοσμίων συνολογών. Έχουμε ανταλλαγή στις υπηρεσίες που ξεπινά τα 700 δις ευρώ ήδη σήμερα. Χωρίς το TTIP σίγουρα μιλάμε για πολύ σημαντικές περιοχές του κόσμου από πλευράς κοινωνικής και οικονομικής. Η ερώτηση είναι εξή. Έναντι τόσο σημαντικού ρόλου που έχουν οι χώρες μας, ε, δεν θεωρείτε ότι όσον αφορά τους Αμερικανούς καταναλωτές, ε, ένα σύστημα ετικετοθεσίας σαφέστερο θα χρειαζόταν ούτω ώστε οι Αμερικανοί καταναλωτέ να, κατα... να, μην συνεχίσουν να καταναλώνουν προϊόντα που θεωρούν ότι είναι ιταλικά ή γαλλικά ή ελληνικά, ενώ στην πραγματικότητα να είναι προϊόντα των ΗΠΑ. Δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να ενώνει τις προσπάθειες που καταβάλουν και η ΕΠΑ και η Ευρώπη. το θέμα των γεγραφικών ενδείξεων είναι καυτό ε, στην Επιτροπή αυτό. Ε, και πιο γενικό ερώτημα αφορά τις μεγάλες καινοτομίες που ε, κάνατε μέσω της τελευταίας ε, νομοσχεδίου ε, της Άμσεν σταματήσατε αντικαταστήσατε με ένα μηχανισμό προστασίας μέσω ασφαλιστικών συστημάτων η ερώτηση είναι πώς έζησαν αυτή την επανάσταση οι Αμερικανοί γεωργοί πρόσφατα μεταρρυθμίσαμε και εμείς την κοινή πολιτική και ίσως σε μερικά χρόνια θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σύστημα. Το θέμα της διαχείρισης των κρίσεων είναι ένα θέμα που συνεχώς βρίσκουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και εγώ σε αυτή την Επιτροπή. Σίγουρα θα ε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Συνάντησα πρόσφατα ε, διάφορους, διάφορα μέλη της ε, Γερουσίας και του Κογκρέσου και κατέστη από τις συζητήσεις ε, εμφανές ότι η Γεωργία στο τέλος ανεξάρτητα από αυτά που θα συζητηθούν στο TTIP θα κάνει τη διαφορά για το TTIP. Θα οδηγήσει επιτυχία ή σε αποτυχία του TTIP η Γεωργία. Κάτι που είναι παρόμοιο και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι ότι αν υπάρχουν γεωργοί δεν θα υπάρχουν τρόφιμα. Αν οι γεωργοί παράγουν τα τρόφιμα, δεν επιτυχάνουν επαρκές εισόδημα, δεν θα υπάρχουν. Οπότε θα έχουμε όλοι προβλήματα. Μεγάλη πρόκληση για μας. Και αυτό που δεν θέλω να γίνει αντικείμενο παζαρέματος ο τομέας της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων στις διαπραγματεύσεις. Ποια είναι η κατάσταση και για τις δύο πλευρές. Όλοι ασχολούμαστε όπως ο κ. Δες με τους τομείς μας. Εγώ θα τα πω στα ράτα. Δεν θέλω να εξαλειφθούν τα κοπάδια των βοηδών στην Ευρώπη. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Δεν θέλω. Θα υπερασπιστώ την κτηνοτροφία. Όπως και από την πλευρά σας. Όλοι έχουμε θέσεις αμυντικές και επιθετικές. Πολλά μπορούν να κερδίσουν όλοι αν καταλήξουμε σε επιτυχή συμφωνία. Κλείνοντας, θέλω να τηρήσω το χρόνο μου. Πιστεύω ότι εάν τα πάμε καλά στο TTIP, θα δημιουργηθούν τεράστια ωφέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρειαστεί χρόνος όμως για τη συμφωνία. δεν θα επιτευχθεί εν μία νυχτή, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν αντιστάσεις στις διαμαρτυρίες. Υπάρχει μεγάλη αντίσταση και παραπληροφόρηση στην Ευρώπη για το τι σε αυτή τη φάση. Χρειαζόμαστε ισορροπημένη, δίκαιη λύση. Και ίσως τα πιο επίμαχα θέματα που αναφέρατε, ίσως θα πρέπει να τα αφήσουμε εκτός για να πετύχουμε τη συμφωνία. Ο κύριος Ρόντε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστώ και για την εισαγωγή και τα ευγενικά σας λόγια για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Συμφωνώ ότι έχουμε μπροστά μας πολύ σοβαρές συζητήσεις ε, εκ μέρου ενό φιλελεύθερου κόμματο, του αδελφού σα κόμματο στην Ευρώπη, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να εντείνουμε τι συζητήσει προκειμένου να διεκπαιρεώσουμε τι διαπραγματεύσει και να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών που θα είναι αμοιβαία υποφελή και για του ε, δύο εταίρου στι δύο όχθε του Ατλαντικού. Οι Αμερικανοί εκτιμούν ιδιαίτερω ε, τα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από αυτή την άποψη όμω έχετε υψηλού δασμού ε, στο βούτυρο και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, οπότε καλό θα ήταν να μειωθούν. Και λυπούμε που το λέω, αλλά είναι δύσκολο να μην αφισβητήσουμε την δέσμευση της ε, Αμερικής για το, ευρωπαϊκό, για το ελεύθερο εμπόριο όταν χτυπά την, ε, τον ευρωπαϊκό γαλακτοκομικό κλάδο με υψηλότερους τους δασμούς στο βούτυρο και την κρέμα γάλακτος. Ευχαριστώ. Η κυρία Σένερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχω τρεις ερωτήσεις. Είπατε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζετε τις μικρομεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Και μάλιστα μιλήσατε για εκμεταλλεύσεις 5, 10, 20 εκταρίων. Ερωτώ λοιπόν, με ποιο μηχανισμό στηρίζετε και προστατεύετε αυτές τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις Επίσης είπατε ότι θέλετε να θρέψετε την ασιατική μεσατάξη. Εγώ φαντάζομαι ότι το ίδιο επιδιώκουν και οι Ασιάτες Γεωργοί. Θέλουν να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν τους πληθυσμούς με τρόφιμα. Οπότε με ποιους μηχανισμούς θέλετε να επιτύχετε αυτό το στόχο σας, τον επισητισμό της ασιατικής μεσαίας τάξης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διαπραγματεύσεις για το TTIP. Είναι διαφανής ο διάλογος που κάνετε, έχει αυτό πρόσβαση η κοινωνία των πολιτών. Επίσης, τι γίνεται για την ποικιλομορφία της Γεωργίας, τι κάνετε και ποια είναι η θέση των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων στη συμφωνία της εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων, το TTIP δηλαδή. Ο κύριος Χόισλενγκ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Γνωρίζετε ότι είναι πραγματικά κρίσιμη συζήτηση στην Ευρώπη για την TTIP. Και οι καταναλωτές συζητούν και οι αγρότες. Πρόσφατα αναθέσαμε μελέτη και από αυτήν βγαίνει ότι θα επωφεληθεί. Τα λέτε εσείς μάλιστα στη δική σας μελέτη, η Αμερικανική Γεωργία, αν μειωθούν οι δασμοί. Άρα δεν μπορούμε να αναμένουμε πάρα πολλά από την TTIP σε ό,τι αφορά την ε, Γεωργία. Έχουμε και το θέμα της ε, τεχνικής των ε, μεταλλαγών. Αντιλαμβάνεστε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν διαφορετική εντύπωση. Το ίδιο για την χρήση ορμονών στην κτηνοτροφία. Κανένα Ευρωπαίο δεν θα πείσετε ότι πρέπει να καταναλώνει κρέας με ορμόνες. Άλλο θέμα που συζητείται εδώ πολύ έντονα είναι η επισήμανση των απογόνων των κλωνοποιημένων ζώων. Κάτι το οποίο απαιτήσαμε εδώ σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με μεγάλη πλειοψηφία. Πώς τα βλέπετε αυτά, είστε διατεθειμένος να δεχτείτε αυτές τις ευρωπαϊκές απαιτήσει. Είπατε ότι όλα αυτά πρέπει να εκτιμηθούν επιστημονικά. Όμως πρέπει να γίνει με σεβασμό και των επιθυμιών των καταναλωτών. Στην επιστήμη μπορούν πολλοί να υποστηρίζουν μια θέση και κάποιοι άλλοι μια αντίθετη θέση. Με τους καταναλωτές τι γίνεται. Μιλήσατε για επισήμανση. Το υποστηρίζω. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρους κανόνες επισήμανσης και ακόμα πιο καθαρή επισήμανση ιδίως σε ό,τι αφορά ε, τους τόπους προέλευσης των προϊόντων. Και να απολούνται και τα τοπικά προϊόντα. Εκεί νομίζω συμφωνούμε. Τέλος έχετε ή έχουμε και συζητήσατε για λίγο ε, για την ε, εταιρική σχέση ή συμφωνία με την άλλη πλευρά του ειρηνικού. Εκεί υπάρχει συμφωνία ότι όντως είναι εποφελής και για τις δύο πλευρές του ειρηνικού. Ακόμα δεν έχει συναυθεί η συμφωνία. Θα περιμένετε να ολοκληρωθεί αυτή πριν να προχωρήσετε με την TTIP στον αγροτικό τομέα. Ο κύριος Άγνιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα σχόλια του κυρίου Νίκολσον. Έχω 7 σύντομα σχόλια. Κυρίως για τα πουλερικά και το κρέας πουλερικών. Καταρχήν, ασφάλεια δικαίου. Στη Βρετανία οι προδιαγραφές μας για τους παραγωγούς ε, και τους εκτροφείς πουλερικών πρέπει να εφαρμόζονται δια νόμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι θέμα διαπραγματεύσεων μεταξύ παραγωγού και πελάτη. Οπότε με αυτό το σενάριο θα ήταν εύκολο οι μεταποιητές στη Βρετανία να, σε, να φέρουν σε δύσκολη θέση τον Βρετανό παραγωγό, να τον υπονομεύσουν. Επίσης, αναφέρατε ότι οι αμερικανικές προδιαγραφές σε θέματα υγείας και ευημερία είναι καλύτερες από τις βρετανικές. Δεν μας πείθετε γι' αυτό. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Τρίτον, αντιβιωτικά. Χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες αντιβιωτικών στην εντατική αμερικανική κτηνοτροφία. Εμείς είμαστε κατά των αντιβιωτικών. Δεν μας αρέσουν τουλάχιστον όχι γενικευμένη χρήση. Μπορείτε να σχολιάσετε αυτό το θέμα της χρήσης αντιβιωτικών. Τρίτο, τέταρτον, χημικά. Εμείς ε, δεν συμφωνούμε με την χημική απολύμαση των σφαγίων. Δεν θεωρούμε ότι είναι ούτε ε, χρήσιμη ούτε αποδεκτή. Επίσης, αυγά από κοδόπουλα ελευθέρας βοσκής. Θα πρέπει να είναι ε, καφέ το τσόφλι τους και να μην έχουν πληθεί, λέμε στη Βρετανία. Ενώ στην Αμερική θα πρέπει να είναι άσπρο το τσόφλι τους και να έχουν πληθεί. Ποιος θα κερδίσει. Γιατί αν κερδίσετε εσείς, τότε θα ε, υπονομευθεί σοβαρότατα ε, ο τομέας μας για τα αυγά από κοντά ελευθέρας βοσκής. Επίσης, για τα απόβλητα. Ένα προϊόν που έχει απαγορευτεί στη Βρετανία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στη, στην, στις Ηνωμένες Πολιτείες τι γίνεται με τα υπόλοιπα των σφαγίων. Χρησιμοποιούνται ως ε, άλευρα και επανέρχονται στην λυσίδα των ζωοτροφών, οπότε τρέφονται τα ζώα με υπόλοιπα σφαγίων. Αυτά, ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον καλεσμένο μας, τον Αμερικανό Υπουργό Γεωργίας, για να δώσει απαντήσεις και θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος ερωτήσεων από τους βουλευτές. Ευχαριστώ. Εκτιμώ ιδιαίτερως την πληθώρα των ερωτήσεων που υποβάλλατε και θα προσπαθήσω να απαντήσω στις περισσότερες. Καταρχήν, από πού πηγαίνουν τα, χρήματα για την υποστήριξη των ε, γεωργών. Αναφέρθηκαν 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Τέσσερα είδη προστασίας και στήριξης δίνουμε. Καταρχήν, ασφάλιση των καλλιεργειών εσωτερική σχέση μεταξύ κυβέρνησης ε, ε, και γεωργών και εξαρτάται το επίπεδο, από τον γεωργό το επίπεδο ασφάλειας που θέλει από την ασφαλιστική εταιρεία. Ένα τμήμα το πληρώνει η κυβέρνηση και αν λάβει χώρα κάποια θεομηνία, ο γεωργός ε, αποζημιώνεται ανάλογα με το είδο κάλυψη που είχε από την ασφαλιστική εταιρεία. Και αν υπάρχει κέρδο από την πώληση αυτών των ασφαλιστικών προϊόντων, το κέρδο το μοιράζονται οι ασφαλιστικέ εταιρείε που διαθέτουν αυτά τα ασφαλιστικά προϊόντα μαζί με την κυβέρνηση. Αν υπάρχουν ζημίε, όπω συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτία ανομβρία εκτεταμένη, και πάλι η κυβέρνηση μοιράζεται με τι ε, ασφαλιστικέ τη εταιρείες της ζημίες. Θέλουμε να προσφέρουμε δέουσα προστασία στου γεωργού, ώστε σε περίπτωση που έχουμε φυσική καταστροφή, κακή καλλιέργεια, κακές μια και να μην πλήττονται. Τώρα, η συμπλήρωση των ασφαλιστικών ε, προγραμμάτων για την καλλιέργεια. Έχουμε διάφορα συστήματα κάλυψη του κινδύνου ή κάλυψη των ζημιών που παρέχουν επικουρική προστασία στους γεωργούς ε, των, της Αμερικής σε περίπτωση που έχουμε κατακόρυφη πτώση των τιμών ε, λόγω ε, θεομηνιών και έτσι εξασφαλίζεται η επιβίωση των γεωργών σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν σοβαρές ε, ζημίες εξαιτία κατακόρυφης πτώσης των τιμών των προϊόντων τους. Πρόσφατα, για παράδειγμα, είχαμε με την γρήπη των πουλερικών ένα πρόβλημα και φυσικά είχε κάτι τέτοιο επιρροή στις τιμές των σιτηρών Γι' αυτό και με βάση αυτά τα δύο προγράμματα στήριξη ε, έλαβαν κάποιο, κάποια αποζημίωση οι γεωργοί γιατί ήταν κάτι απρόβλεπτο και κάτι που εξέφευγε από τον έλεγχό του. Βέβαια δεν ε, μπόρεσαν να υποφεληθούν από θέματα ασφάλεια των καλλιεργειών, γιατί η κάλυψη τέτοια προβλέπεται μόνο σε περίπτωση αμυνία και όχι όπω είχαμε την περίπτωση τη επιζωτία τη γρήπη. Επίσης, ε, δίνουμε τους ε, γεωργούς να ασχολούνται με τη συντήρηση του εδάφους και σε ό,τι αφορά την κτηνοτροφία, με εξαίρεση τα πουλερικά, την κτηνοτροφία, εκεί έχουμε πρόγραμμα καταστροφών και αν λόγω ε, ξηρασία χαθούν ζωοτροφέ, υπάρχει θεομηνία ή καταιγίδα ή ένα σοβαρό πρόβλημα που οδηγεί σε απώλεια του, των πουλερικών, τότε υπάρχει ένα, πρόβλημα, ένα πρόγραμμα παροχής βοήθειας. Αξαρτάται από τι θα συμβεί. Έχουμε λοιπόν τέσσερα είδη στήριξη που παρέχουμε στου γεωργού και κτηνοτρόφου. Και υπάρχουν και πολλά άλλα προγράμματα, αλλά νομίζω ότι αυτά ήταν τα βασικά που δίνουν μια ιδέα για το πώ στηρίζουμε του γεωργού και κτηνοτρόφου μα. Το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων είναι πολύ σοβαρό θέμα. Υπάρχουν κάποιοι όροι, υπάρχουν κάποιοι δείκτες που καθορίζουν τα προϊόντα και που είναι τόσο γενικοί και χρησιμοποιούνται τόσο ευρέως που θα ήταν δύσκολο να έχουμε να καταλάβουν οι Αμερικανοί καταναλωτές μια αλλαγή του συστήματος για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Γι' αυτό είπαμε καλό θα ήταν υπάρχει μια διαδικασία παροχής σήματος ώστε όσοι θέλουν να προστατεύσουν ένα προϊόν από συγκεκριμένη περιοχή της Ευρώπης να το κάνουν με ένα συγκεκριμένο σήμα. Για παράδειγμα συγκεκριμένα τυριά. Θα μπορούσαμε με εμπορικά σήματα συγκεκριμένα που θα δίνονται στους παραγωγούς ε, συγκεκριμένων τύπων τυριών όταν φτάνουν αυτά τα τυριά στις αγορές μας θα ξέρουν οι καταναλωτές μας ότι τα συγκεκριμένα τυριά τα αγοράζουν από την Ιταλία, αυτά προέρχονται από την Ιταλία. Φυσικά αυτό θα το συζητήσουμε περαιτέρω στις διαπραγματεύσεις, το θέμα των γεωγραφικών αδείξεων και σίγουρα δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε λύση. Πάντως, αν έχουμε χρόνο και καλή επικοινωνία μεταξύ μας, θα καταφέρουμε να προσπίσουμε τα συμφέροντα όσων υπέρ τέτοιων προτάσεων που έχουν προστιθέμενη αξία, χωρίς να φέρουμε σε δύσκολη θέση τους Γεωργούς, είτε τους Αμερικανούς, είτε τους Ευρωπαίους και να μην διακυβεύουμε την επιβίωσή τους. Επίσης, είπατε πώς αντιδρούν στον νέο νόμο οι Αμερικανοί γεωργοί. Εκτιμούν ιδιαίτερα στο γεγονό ότι ο νέο γεωργικό νόμο ε, προβλέπει αυτά τα, τα προγράμματα προστασία από τι ομιλίε, κάλυψη ασφαλιστική ε, και συντήρηση και μάλιστα πέρυσι είχαμε την καλύτερη εφαρμογή. Και είναι τελευταίο γεωργικό νόμο σε μια σειρά 6-7 και ήταν ο πιο επιτυχημένο. Επίση έχουμε το πρόγραμμα προστασία για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, για του γαλακτοπαραγωγού που μπορούν να αγοράσουν σε ένα επίπεδο ασφάλειας ε, κατά των ε, πολύ χαμηλών τιμών. Και όταν η διαφορά μεταξύ των της τιμής των και της ε, τιμής του γάλακτος πέφτει, τότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός. Το θέμα είναι αν είναι ικανοποιημένη η γαλακτοπαραγωγή, γιατί υπάρχουν διαφορές στις των τροφών μεταξύ των διαφόρων πολιτιών. Αυτό ίσω δεν λαμβάνεται υπόψη από τον γεωργικό νόμο και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί στη συνέχεια. Πάντω, γενικώ, η γεωργία είναι σχετικά ικανοποιημένη με τι μεταρρυθμίσει του νέου γεωργικού νόμου. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, η γεωργία σίγουρα είναι το τελευταίο θέμα που ε, εξετάζεται σε μια εμπορική συμφωνία και το TTIP δεν αποτελεί εξαίρεση. Το γαλακτοκομικό θέμα, ο γαλακτοκομικό στο ήταν το τελευταίο θέμα στι συζητήσει. Πάντω ε, ελπίζω ότι για πολύ καιρό θα ασχοληθούμε και με τα γεωργικά θέματα στα πλαίσια του TTIP. Τώρα, ακριβώς επειδή η γεωργία καλύπτει για ένα θέμα καλλιέργειας, δεν είναι μόνο η παραγωγή ενός τροφίμου, αλλά είναι ένα θέμα ολόκληρης νοοτροπίας, ολόκληρης γεωργικής παιδείας και κουλτούρας. Το θέμα της κουλτούρας είναι πολύ σημαντικό γιατί σε κάθε χώρα οι γεωργοί ταυτίζονται με τις καλλιέργειές τους. Είναι θέμα προσωπικό και θέμα ταυτότητας. Τώρα, για μας η πρόκληση είναι ότι η γεωργία δεν είναι τόσο μείζον πολιτικό ζήτημα ώστε να περάσει σε μια συμφωνία. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά σοβαρό πολιτικό θέμα για να σταματήσει μια συμφωνία. Οπότε εδώ ιδέουσα προσοχή στη γεωργία ή στα γεωργικά συμφέροντα σε μια εμπορική συμφωνία πολύ συχνά δύσκολα περνάνε και περαιώνει τη διαδικασία για τι εμπορικέ συμφωνίε. Για παράδειγμα, αν είχαμε μια συμφωνία TTIP χωρί τη γεωργία, που θα παραμέριζε τη γεωργία επειδή θα ήταν δυσεπίλητη η συμφωνία για το γεωρικό θέμα, πολύ δύσκολα θα συγκέντρωνε στο Κογκρέσο συμφωνία για να κυρωθεί. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα δύσκολα αυτά, τις επίλυτα γεωρικά θέματα, παρόλα αυτά να τα περιλάβουμε στην TTIP. Τώρα, για τους γεωργούς. Φυσικά, αν σταματήσουν οι γεωργοί να δουλεύουν, δεν θα έχουμε εμείς τρόφιμα και θα είστε και πολλοί από εσά ε, γεωργοί. Οι υπόλοιποι όμως ε, που δεν είμαστε γεωργοί έχουμε εκχωρήσει την ευθύνη του επιστησμού της ε, τροφοδοσίας των οικογενειών μας στους γεωργούς. Γιατί άλλος είναι δικηγόρος, εγώ είμαι δικηγόρος, η γυναίκα μου καθηγήτρια. Ο καθένας λοιπόν επιδίωξε το όνειρό του, το ίδιο θα κάνουν και τα παιδιά μας, αλλά δεν έχουμε δεν είχαμε εμπειρία με τα γεωργικά θέματα. Και ακριβώ καταφέραμε εμεί να υλοποιήσουμε τα όνειρά μα, επειδή χωρίσαμε το θέμα τη παραγωγή τροφίμων στου γεωργού. Και είναι σημαντικό να του αναγνωρίσουμε τη σημαντική του συμβολή, γιατί μερικέ φορέ παραγνωρίζεται η σημαντική συμβολή τη γεωργία. Και μάλιστα στην πατρίδα μου το κόστο των τροφίμων είναι σχετικά χαμηλό. Είναι ένα τμήμα του προπολογισμού του νοικοκυριού. Αφιερώνεται ένα τμήμα του μισθού μας στην αγορά τροφίμων. Γι' αυτό και πολλοί θεωρούν ότι υπάρχουν ε, ε, και υπάρχει και μεγάλη διαθεσιμότητα, υπάρχουν και πιστιστικά προγράμματα. Γι' αυτό δεν εκτιμούν, ο κόσμο δεν εκτιμά ιδιαίτερω ίσω την αξία τη γεωργία και των τροφίμων. Και χαίρομαι που εμεί το τονίζουμε αυτό ιδιαίτερο. Τώρα υπάρχουν πολλά σχόλια που μιλάνε για τι διαφορετικέ μεθόδου παραγωγή μεταξύ Αμερική και Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, χρήση ορμονών ή μέθοδοι φτηνοτροφίας που είναι διαφορετικές στις διόχθες του Ατλαντικού. Πάντως ε, οι καταναλωτές είναι έξυπνοι, ξέρουν τι θέλουν και είναι ικανοί να κάνουν τις σωστές επιλογές. Και αν μια αγορά είναι ανοιχτή και εγώ προσπαθήσω να πουλήσω κάτι που ο Ευρωπαίος καταναλωτής ε, δεν θέλει να το αγοράζει, τότε εγώ κατά πάσα πιθανότητα θα σταματήσω να προσπαθώ να το πουλάω στην αγορά ή θα χρειαστεί να αλλάξω το προϊόν μου αν θέλω να το διαθέσω. Νομίζω ότι αυτή είναι μια φυσιολογική εξέλιξη που είναι συναφής και με τη φύση του αγορά. Καλύτερα την επιλογή να την κάνει ο τελικός καταναλωτής και όχι η κυβέρνηση σε προγενέστερο επίπεδο. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει βέβαια ένα επίπεδο διαφάνειας και σωστή ενημέρωση των καταναλωτών ώστε τεκμηριωμένα να, να κάνουν τις επιλογές τους. Και σίγουρα θα εξετάσουμε αυτό το θέμα πιο διεξοδικά για να δούμε πώς θα ενημερώνουμε διόντως τους καταναλωτές μας ώστε έχοντας γνώση να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους. Το θέμα του βουτύρου. 150% ήταν η αύξηση στις εισαγωγές ε, ευρωπαϊκού βουτύρου στην Ευρωπαϊκή, στην, ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και με βάση τα δικαιώματά μας στον ΠΟΕ επιβάλαμε ένα επίπεδο δασμού που είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό που επιτρέπει ο ΠΟΕ και εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Κατά μια προσπάθεια για να ανταποκριθούμε σε μια πολύ σημαντική και άνευ προηγουμένου για πολύ καιρό αύξηση των εισαγωγών βουτύρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως ε, την ανησυχία σας ε, μου τη μεταβίβασε πολλές φορές και ο Επίτροπος Χόγκαν. Επαναλαμβάνω, το μέτρο αυτό της αύξησης των δασμών ε, είναι περιορισμένο και ως προς το πεδίο εφαρμογή, την ευέλεια του και χρονικά περιορισμένο. Τώρα, πώς στηρίζουμε τους μικρομεσαίους γεωργούς. Έχουμε ένα πρόγραμμα «Μάθε τον γεωργό σου». Έχουμε ένα πρόγραμμα μικροδανείων με δάνεια προς, μικρά δάνεια προς τους γεωργούς σε μικρές εκμεταλλεύσεις Έχουμε και ένα πρόγραμμα συντήρησης ώστε η καλλιεργητική περίοδος να παραταθεί με θερμοκήπια. Παρέχουμε συνδρομή στα, με ιδιαίτερες πληροφορίες για τη θέση εμπορία και ε, τις τιμές για να ξέρουν οι γεωργοί πώς μπορούν να διαθέσουν καλύτερα το προϊόν τους και σε τι τιμές. Προωθούμε τα τοπικά προϊόντα και επίσης ε, προωθούμε συνεργασία των τόπιων γεωργών με τα σχολεία. Είχαμε 220 επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις σε ε, σχολεία και 6,5 εκατομμύρια μαθητές επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα αυτό. Μία ενημέρωση των μαθητών για τη γεωργία, για το πώς γίνεται η παραγωγή, η καλλιέργεια και έτσι προωθούμε τους μικρούς γεωργούς, τους μικρούς παραγωγούς. Βέβαια, οι μικροί παραγωγοί ε, τα βρίσκουν σκούρα σε μια αγορά βασικών προϊόντων που επιβραβεύει κυρίω την αποτελεσματικότητα και την τεχνολογία. Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε μια διαδικασία όπου και οι μικροί παραγωγοί και οι τόπιοι παραγωγοί να έχουν προσωπικέ σχέσει και επαφέ με του πελάτε, γιατί μπορεί ο πελάτη να θέλει να πληρώσει και λίγο ακριβότερα το προϊόν, ακριβώ επειδή γνωρίζει, αυτή, γνωρίζει τον Γιώργο, εκτιμά αυτή την διαπροσωπική σχέση, ξέρει την προέλευση του τροφίμου και αυτό είναι διατεθειμένο να το πληρώσει και λίγο ακριβότερα. Οπότε, αν μπορέσουμε να στηρίξουμε, έτσι μπορούμε να στηρίξουμε και την ποικιλομορφία και την πολυμορφία της Αμερικανικής Γεωργίας. Σε ό,τι αφορά το TPP, την ε, Συμφωνία του Ειρηνικού και την Ασιατική Μεσαία Τάξη, γενικώ πιστεύω ότι θα αυξηθούν οι επιστηστικές ανάγκες ε, αισθητά. Και με τους σημερινούς αριθμούς δεν θα καταφέρουμε να θρέψουμε τον κόσμο στο μέλλον. Ούτε καν την ασιατική μεσαία τάξη στο μέλλον. Την περασμένη εβδομάδα πήγα στην Κίνα και 10 εκατομμύρια γεωργοί εγκαταλείπουν τις ε, καλλιέργειές τους κάθε χρόνο. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα γιατί δημιουργεί τεράστιε κοινωνικέ προκλήσει. Πάντω αναγνωρίζουν οι Κινέζοι ότι αυτή τη στιγμή η γεωργία του δεν ανταποκρίνεται στι ανάγκε του πληθυσμού. Γιατί ο πληθυσμό αυξάνεται και η γεωργία δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την αύξηση, τη δημογραφική. Ε, παρόμοιες ε, έχουμε και τη Μαλαισία, το Βιετνάμ, την Κορέα, την Ιαπωνία και όλοι αναγνωρίζουν τι προκλήσει θα δημιουργηθούν τεράστιες επιχειρηματικές ε, ευκαιρίες στη γεωργία για όλους και αυτό δεν σημαίνει ότι ε, θέλω να πουλήσω στην Ασία εις βάρος των, γεωργών, των ε, Ευρωπαίων γεωργών. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή δουλειά για όλους στο εγγύς κυρίως ό,τι αφορά την παραγωγή πρωτεϊνών, γιατί θα υπάρξει τεράστια αύξηση στη ζήτηση των πρωτεϊνών και ταυτόχρονα θα έχουμε και την αλλαγή του κλίματος. Θα δούμε τι προϊόντα θα καλλιεργούνται, σε τι επίπεδο, γιατί θα αλλάξουν και οι εποχές της καλλιέργειας, η διάρκειά τους, γιατί σήμερα μπορεί να καλλιεργούμε κάπου καλαμπόκι, αλλά σε τέσσερα χρόνια δεν είναι σίγουρο ότι θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Θα γίνουν πολλές αλλαγές εξαιτία των κλιματικών αλλαγών, θα γίνουν αλλαγές και στη γεωργία. Γι' αυτό και θέλουμε να εφοδιάσουμε τους γεωργούς μας με στρατηγικές προσαρμογής και κατευνασμού των συνθήκων, μετριασμού των συνθήκων και των κλιματικών αλλαγών. Τώρα για τη διαφάνεια. Πρόσφατα είχαμε ε, το νόμο για την εμπορική αρχή που προβλέπει ότι κάθε εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύεται η διοίκηση θα πρέπει να τίθεται στο διαδίκτυο και να είναι προσιτή στο κενό για αρκετό διάστημα και νομίζω ότι αυτό εξασφαλίζει διαφάνεια και αυτές οι εμπορικέ συμφωνίες θα, βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων για πολύ καιρό, γιατί είναι χιλιάδες οι σελίδες τη Εμπορική Συμφωνία και του ειρηνικού. Φαντάζομαι το TTIP θα είναι αντίστοιχο ογκώδες έργο και μακροχρόνιες θα είναι και συνέπειε, Γι' αυτό και θέλουμε διαφάνεια και θα την εξασφαλίσουμε, τουλάχιστον στι Ηνωμένε Πολιτείε θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος σε όλους τους ενδιαφερομένους για να κάνουν τις επιλογές τους. Τώρα, αναφέρθηκε το θέμα της μικροβιακής αντίστασης, μικροβιακής αντοχής. Εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα προκειμένου να μειώσουμε αισθητά τη χρήση των αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία. Συνεργαζόμαστε με κτηνιάτρους για θέματα μικροβιοικής αντοχής και να μην, αποφασίσαμε να μην χρησιμοποιούμε ε, τα αντιβιωτικά ως μέσα ως ανάπτυξη, αλλά μόνο για θεραπεία. Ε, θέλουμε να καταλάβουμε πώς δημιουργείται αυτή η μικροβιακή αντοχή και γι' αυτό έχουμε συντονισμένες προσπάθειες μεταξύ των γιατρών και των κτηνιάτρων, ώστε να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση υγειονομική στο θέμα αυτό. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα υπάρχει μια ειδική μονάδα στην κυβέρνηση που συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας για το θέμα αυτό. Αναφέρθηκαν τα μεταλλαγμένα, οι ορμόνες, οι γεωρικές ενδείξεις και το πώς θα ζητηθούν στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης TTIP και το πώς θα λιάνουμε τις διαφορές μεταξύ μας. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολες οι διαπραγματεύσεις, δεν έχουμε αυταπάτες, θα είναι δύσκολες, επίπονες, θα απαιτήσουν χρόνο, θα απαιτήσουν δέσμευση και διάθεση να βρούμε μια αμοιβαίως υποφερή λύση και φυσικά θα πρέπει να έχουμε αμοιβαία κατανόηση των συστημάτων μας, των στόχων μας και θα χρειαστεί και κάποια δημιουργικότητα και ευρηματικότητα, ώστε να καταλήξουμε σε ένα λειτουργικό σύστημα. Γιατί η εμπειρία μας και η ιστορία έχει δείξει ότι τέτοιες εμπορικές συμφωνίες ε, δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα μία χώρα να υποφέλει της βάρος άλλης. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο ούτε στη Γεωργία, ούτε στο TTIP, ούτε στην Συμφωνία του Ειρηνικού. Θα πρέπει να είναι αμοιβαία υποφελή συμφωνία, γιατί αν ωφελεί μόνο το ένα μέρος, τότε είναι αποτυχημένη. Μία στιβαρή εμπορική συμφωνία είναι μια συμφωνία που δίνει την ευκαιρία σε όλους τους συμβαλωμένους να είναι αποτελεσματική και ταυτόχρονα δίνει ένα ευρύ φάσμα επιλογών στους καταναλωτές. Δίνει ποικιλία ε, σε χαμηλότερο κόστος και θα πρέπει να βρούμε όλοι δημιουργικού και ευρηματικού τρόπους να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας. Αυτά θα είναι τα ωφέλη και τα προτερήματα μιας σωστή εμπορικής συμφωνία. Και αυτές τι φιλοδοξίε έχουμε και από το TTIP. Και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Αυτή τη στιγμή συζητάμε το θέμα της σήμανσης, της ετικετοθεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρότεινα ε, να μην έχουμε παλαιομοδίτικε συζητήσει, συζητήσει τύπου 20ου αιώνα για τον 21ο αιώνα. Θέλουμε πιο καινοτόμε συζητήσει, γιατί έχουμε όλο και περισσότερου με κινητά που έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία την ε, αξιοποιούνται και την αξιοποιούνται όντω. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γραμματού ε, κωδικού και να μπορούν οι καταναλωτέ να κάνουν τι επιλογέ του έχοντα γνώση τη κατάσταση. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τι νέε τεχνολογίε με σωστά μηνύματα και για την ασφάλεια και για την ε, βιωσιμότητα του προϊόντο. Γιατί είδαμε ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα δεν ε, ε, ενέχουν κινδύνους για την υγεία. Παρόλο που μερικοί διαφωνούν, οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί. Οπότε θα πρέπει τις πληροφορίες να φτάνουν στο καταναλωτή με τρόπο που δεν θα δίνει λάθος μηνύματα για την ασφάλεια ενός προϊόντος. Επίσης έχουμε σήμα για τη διατροφή ή για την έλλειψη κινδύνου. Τέτοιες πληροφορίες θέλουν οι καταναλωτές. Θρεπτική αξία και έλλειψη κινδύνου. Έτσι μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στο μανάβικο, να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να κάνει την επιλογή του έχοντας γνώση της κατάστασης. Σωστή ενημέρωση είναι παρα, απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνουν σωστές επιλογές οι καταναλωτές. Τώρα το θέμα της σπαγκώδης εγκεφαλοπάθειας, BSC. Φυσικά μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα και ήμασταν πολύ επιθετικοί στις προσπάθειές μας να αποτρέψουμε ε, να συμπεριλαμβάνονται στις ζωτροφές... Ε, ύποπτα συστατικά που θα ενισχύει τον κίνδυνο για εμφάνιση της, βόδους, ε, της ε, εγκεφαλοπάθειας των βοηθών, της πονκόδους εγκεφαλοπάθειας. Οπότε τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά κατά τη γνώμη του ελάχιστον δεν είναι ανυπέρβλητα. Και το θέμα των αυγών από κότες ελευθέρας φωσκής, και εκεί μπορούμε να, να τα βρούμε να μπορούν οι καταναλωτές που θέλουν καφέ, αυγά, αυγά με καφέ τσόφλι να τα αγοράζουν, το ίδιο καφέ που θέλουν αυγά με λευκό τσόφλι να μπορούν να τα αγοράζουν. Δεν νομίζω ότι θα είναι αδύνατο να καταλήξουμε στη συμφωνία σε αυτά τα θέματα. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο απαντήσεων και περνάμε στο δεύτερο με τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Παρακαλώ ένα λεπτό καθένας και να σεβαστείτε το χρόνο σας και να αποφεύγετε τις επαναλήψεις. Νομίζω το απαιτεί η ευγένεια να είμαστε συνοπτικοί. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Υπουργέ για τον χρόνο σας. Μία συγκεκριμένη ερώτηση για την συμφωνία TTIP για τις ε, ρυθμίσεις SPS και στην ε, και στι Ηνωμένε Πολιτείες έχετε μεγάλο πρόβλημα να δείτε την Ευρώπη σαν ένα σύνολο. Και πολλές ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν να είναι δίθεν ένα συνονθήλευμα 28 χωρών μελών, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθμίζεται με κανονισμούς και οδηγίες. Αλλά βεβαίως την ευθύνη της εφαρμογής τους φέρουν οι χώρε μέλη. Μα το ίδιο συμβαίνει και στι ΗΠΑ. Οι επιμέρου πολιτείε σα φέρουν την ευθύνη εφαρμογή των ομοσπονδιακών νόμων. Στην, ε, Αμερική, στην Ευρώπη, συγγνώμη, ποτέ δεν θα ε, είχαμε τέτοια εντύπωση. Πώ τα βλέπετε λοιπόν και πώ μπορούμε, πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Ε, Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι μεγάλο κομμάτι της αγοράς αφορά προϊόντα προστατευμένα. Πώς θα αποφευθούν τα παραποιημένα προϊόντα, η διάθεσή τους στην αγορά, Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα γι' αυτό. Δεύτερο. Πρέπει να πω ότι για την Ουγγαρία όσον αφορά τη διαθέτηση των διαφορών Φοβόμαστε την επεξεργασία των πουλερικών με χλωρίνη ή γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ας πούμε ότι θα απαγορευθούν στην Ουγγαρία. Φοβόμαστε όμως ότι τότε θα καταβάλουμε κάποια πρόστιμα. Πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Κύριε Σαντριέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και εσάς κύριε Υπουργέ για αυτά που είπατε. Άκουσα και βλέπω πόσο υπάρχει απόσταση μεταξύ των προσεγγίσεών σας και των δικών μας. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο TTIP και συγκεκριμένα θέματα. Να εμβαθύνουμε κάπου. Ο ενδέκατος γύρος των συζητήσεων τον Οκτώβριο ε, μας οδήγησε κάποιες φορές δασμολογικές και ξέρω ότι πραγματικά η γεωργία μας θα ευνοηθεί από την ελάφρυνση από τους τασμούς εάν οι μη τα μη δεσμολογικά εμπόδια φυτογενομικά μη φυτογενομικά αρθούν. Και αυτό ε, και ένα σημείο είναι και αυτό η αναγνώριση της προστασίας των ε, γεωγραφικών ενδείξεων των ευρωπαϊκών. Είναι κάτι απαραίτητο για μας να για να υιοθετηθεί συμφωνία. Θα ήθελα να σας ακούσω πάνω σε αυτό. Ποια ακριβή προβλήματα δημιουργούν οι γεωγραφικές ενδείξεις σήμερα για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ερένς Γκαρσία. Eh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Έχω δύο ερωτήσεις. Δεν θεωρείτε κύριε Υπουργέ ότι θα ήταν χρήσιμο στην Ευρώπη να έχουμε νομοθεσία παρόμοια με αυτή που έχει η Αμερική και η FDA για την επισητιστική άμυνα. Γιατί μόνο προαιρετικά τέτοια μέτρα έχουμε και κυρίως είναι ιδιωτική υφή. Δεν υπάρχει τέτοια κοινοτική ή κρατική νομοθεσία. Δεύτερον, δεν θεωρείτε ότι μου θα ήταν να κάνετε μια χειρονομία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας άμεσα τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα, τις, ε, ε, τα POP, τις ονομασίες προέλευσης γιατί έτσι θα μας βοηθούσε πολύ να προχωρήσουμε στη διαπραγματεύσεις του TTIP. Γιατί δεν χρειάζεται ε, να έχει κανείς διπλωμά τεχνίας για να ε, δίνει, ε, για να παράγει τυρί από το πιαμόντε. Γιατί το πιαμόντε είναι μόνο στην Ιταλία. Το ίδιο συμβαίνει με κρασί της Μάλαγας ή από τη Μάλαγα ή μεταξύ από το Χερές ή από ένα προϊόν που μπορεί να έχει συγκεκριμένη ονομασία από τη Γερμανία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι Ιρλανδός βουλευτής κύριε Υπουργέ. Έχω δύο ερωτήσεις που σχετίζονται με το Βόιο. Πρώτον, διαπραγματεύσεις TTIP. Η ΕΠΑ έχει 45.000 τόνους αδοσμολόγητο όριο ποσόστοση για βόιο χωρίς ορμόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να αναφερθείτε στη διαπραγματευτική σας θέση σε ποιο ύψος θέλετε να φτάσει αυτός ο αριθμός όσον αφορά το βόιο το, από ΕΥΠΑ που θα μπαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεύτερο ερώτημα. Ίσως στην Ιρλανδία επανειλημμένα. Και υπογραμμίστηκε ότι θα ανοιχτεί στο Ιρλανδικό βόιο τότε η Αμερικανική αγορά και τότε ο υπουργό μας και οι ομολογοί του της ΙΠΑ εκτιμούσαν ότι η αγορά των ΙΠΑ θα άξιζε 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τους Ιρλανδούς παραγωγού βοήου. Φέτο το πρώτο εξάμεινο όμως οι εξαγωγέ από την Ιρλανδία στη ΣΥΠΑ του βοήου ήταν 194.000 ευρώ. Γιατί αυτό το στοιχείο, αυτός ο αριθμός είναι τόσο χαμηλό, θα αυξηθεί? Και τι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί σημαντικά αυτό το ποσό, κυρία, κυρία Μίλλερ. Προέρχομαι από μια μικρή ορεινή περιοχή, κύριε Υπουργέ, με μικρές παραγωγές τυριού κυρίως, με γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης. Και είμαι πεπισμένη ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας θα χάσουν αν εφαρμοστεί, αν ψηφιστεί, δηλαδή συναυθεί και εφαρμοστεί η TTIP. Σε συζητήσεις με την Επίτροπο που είναι αρμόδια για ζήτηματα εμπορίου ακούμε ότι από τους Αμερικανούς δεν φαίνεται να γίνεται προσέγγιση προς τις ευρωπαϊκές θέσεις, δηλαδή για θέματα γεωργικά. Και εσείς πολύ λίγα είπατε σε ό,τι αφορά την κλωνοποίηση. Μέσα εδώ στην Ευρώπη δεν την θέλουμε την τεχνολογία αυτή. Θα ήθελα να ακούσω από εσά εάν επισημαίνετε τα τρόφιμά σας, εάν είναι ξεκάθαρη η επισήμανση αυτή ή αν μόνο τα γράφετε αυτά στα βιβλία που τηρούν οι εκτινοτρόφοι και θέλω να γνωρίζω και πόσοι γεωργοί παροιμήν, σαν δηλαδή, παράγουν βιολογικά προϊόντα. Παίζουν κάποιο ρόλο τα πράγματα αυτά. Γιατί εμείς εδώ συζητούμε για την προστασία των ζώων, ευημερία των ζώων και αυτά νομίζω ότι όλα έρχονται σε αντίθεση τελικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία TTIP. Ο κύριος Χάιτεμα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Υπουργό που ήρθε. Μας ενδιαφέρει ο γεωργικός σας νόμος. Ο τελευταίος γεωργικός νόμος αναφέρεται περισσότερο στην διαχείριση κινδύνου. Γιατί? Γιατί αλλάξει η πολιτική σας ως προς αυτό το σημείο και πώς επηρέασε και τον προϋπολογισμό αυτή η αλλαγή. Ε, δαπανάτε περισσότερα κονδύλια για την έρευνα, την καινοτομία, όχι μόνο για την ακριβή γεωργία, αλλά και την έρευνα για την ποιότητα του εδάφους και το καθεξής. Επίσης, στην Συμφωνία του Ειρηνικού, που πού βρέθηκαν οι σκόπελοι και πώς μπορούμε τα διδάγματα της Συμφωνίας του Ειρηνικού να τα αξιοποιήσουμε στο TTIP. Κύριε Σάιερ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Σάιερ. Διαπιστώνω μια θετική ε, προσέγγιση από μέρους σας. Εμείς από τις κατοχώρες δηλαδή, σε ό,τι αφορά προκυπευτικά... χειροτροφία και εκτινοτροφία γενικότερα, τηρούμε πάντοτε κριτική στάση και δεν θέλουμε την TTIP. Εσείς φαίνεται όμως να ε, ενδιαφέρεστε και για τις ε, αγροτικές οικογένειες και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Πράγματα που και αποχρώσεις που δεν έχουμε ακούσει ποτέ από την Κίνα για παράδειγμα. Έγινε εδώ και μεγάλη διαδήλωση στις Βρυξέλλες μάλιστα πρόσφατα αγροτών με μέλη και αγροτικών οικογενειών τι γίνεται με τον ανταγωνισμό οι αγρότες θέλουμε εμείς να έχουν ένα επαρκές εισόδημα. Αν μπορούμε με συνεργασία Ευρωπαίοι και Αμερικανοί να εξασφαλίσουμε ένα καλό εισόδημα του γεωργός, τότε ίσως να συμφωνήσουμε και στην TTIP. Εφτά δισεκατομμύρια είμαστε οι άνθρωποι στον κόσμο, ενώ ήμασταν 3,5 το 1970. Άρα με όσα επιτύχαμε ως τώρα με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κτλ. δεν καταφέρουμε να τους θέσουμε όλους αυτούς. Και η παραγωγή υφίσταται τα δεινά. Βεβαίως και είναι ρεαλιστές οι Αμερικανοί και βέβαια και βλέπω και το αγροτικό σας νομοθέτημα, Farm Bill, την προστασία απέναντι στους κινδύνους, την προστασία του εισοδήματος κτλ. Μεγάλες οι διαφορές. Εσείς ε, τις ενισχύσεις τις λέτε κοινωνικές ενισχύσεις και μπαίνουν στο πράσινο καλάθι του, ε, του ΠΟΕ. Γι' αυτό φοβούμαι εγώ πολύ την συμφωνία της ΤΥΠ. Είπατε και ο ίδιος ότι η γεωργία είναι και το τελευταίο, ε, η τελευταία πτυχή της ΤΥΠ. Αλλά μπορεί αυτή να ρίξει ολόκληρη τη συμφωνία. Τώρα για το βοδινό. Είπατε ότι θα έχουμε παρόμοια συστήματα. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή θα έχουμε ε, κανόνες ή και θα γίνει προσπάθεια ευρωγνωμών να συγκλίνουν. Καπούτο. Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζω με μεγάλη χαρά τον Αμερικανό Υπουργό Γεωργίας. Μεγάλη τιμή για αυτή την Επιτροπή να τον υποδέχεται εδώ σήμερα. Ερώτηση που θέλω να θέσω. Ίσως ήδη έχει κάπως καλυφθεί, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διευκρίνηση. Αναφερθήκατε ότι δεν μπορούμε να έχουμε, στο δεν μπορούμε να έχουμε δύο ίδιες ίσες αγορές. Πρέπει να έχουμε αντίστοιχα συστήματα, όχι ταυτόσημα. Ε, και αναφερθήκατε σε κάποια ζητήματα βασικά, όπως και την αρχή της πρόληψης που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη, και την προσέγγιση με την εξακρίβωση του κινδύνου, την αποτίμηση του κινδύνου στη ΣΥΠΑ. Μετά είναι και το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων. Το Wall Street Journal έλεγε στην επικεφαλή τι είναι πιο αμερικάνικο από το τυρί παρμεζάνο, έλεγε. Εκεί βλέπουμε τη διαφορά της προσέγγισης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ερώτησή μου. Στην παρέμβασή σας τονίσατε την ανάγκη αντιστοιχεία γεωγραφικών ενδείξεων με το σήμα. Γιατί να μην υπάρχει αυτοματισμός που θα αναγνωρίζει στις γεωγραφικές ενδείξεις αυτομάτως έναν ορισμό σήματος που θα παίρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, συγγνώμη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Μιλήσατε για τις διαφορές μεταξύ της Αμερικανικής και της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι οι ευρωπαϊκές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι 10 φορές μικρότερες κατά μέσο όρο από τις αμερικανικές. Επίσης, ε, διαφορετική τεχνολογία χρησιμοποιούμε, διαφορετική αντιμετώπιση των αντιβιωτικών, των ορμονών που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ εμείς ε, επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη πέθρου, σε μια φιλοπεριβαλλοντική καλλιέργεια, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παρεμβαίνουν μόνο σε θέματα αγοράς και μόνο σε περίπτωση θεομηνιών. Με βάση όλες αυτές τις διαφορές, πιστεύετε ότι είναι δυνατόν σε μια εμπορική συμφωνία να έχουμε ένα νέο πλαίσιο που θα λιένει αυτές τις διαφορές και θα μας επιτρέψει να φτάσουμε σε κάποια σύγκληση. Εμείς εκπροσωπούμε μια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών αμφιβάλλω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σύγκληση απόψεων τελικά. Ο κύριος Χόιμπους, η κυρία Χόιμπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Υπουργέ. Ερώτηση για, νόε, για νέες τεχνολογίες ε, στην κτηνοτροφία. Συν, συναντηθήκατε με εκπροσώπους των επιχειρήσεων γενετικής τεχνολογίας που ζητούν να μην ρυθμίζονται, να μην ομοθετούνται δηλαδή τα της χρήσης γενετικής τεχνολογίας όπως γίνεται και στη Νέα Ζηλανδία. Στις ΗΠΑ τι προτίθεται να κάνετε. Είπατε ότι είναι ξύπνοι οι καταναλωτές και μπορούν να διαλέξουν μόνοι τους. Οι πληροφορίες όμως που δίνονται στην, ε, στις ΗΠΑ δεν αναφέρονται στη γενετική τεχνολογία που εμπεριέχεται στο προϊόν. Ενώ στην Ευρώπη ναι. Και είπατε ακόμη ότι αυξάνονται οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις στις ΗΠΑ. Ακόμα και αν χρησιμοποιούν όμως γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Πώς θα προστατεύσετε τις βιολογικές σας εκμεταλλεύσεις από την μετάδοση των ε, γενεολογικά ε, τροποποιημένων οργανισμών, ενώ εμείς εδώ ζητούμε μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτούς. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας πιστεύω κύριε Υπουργέ ότι φροντίζετε για τα δικαιώματα και την υγεία των καταναλωτών όπως και εμείς ε, κάνουμε το ίδιο και τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Αλλά όπως είπατε έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις σε πολλά θέματα και διαφορετικές προδιαγραφές. Γι' αυτό έχουμε και πολλά έκρεμη θέματα, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι στη Γεωργία. Η Αμερικανική νομοθεσία είναι αρκετά φιλελεύθερη και ανοιχτή και ανέχεται και χωρίς μάλιστα σήμανση την παρουσία γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στα τρόφιμα. Ενώ οι δικοί μας καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν τι τρώνε. Οπότε, στον τομέα αυτό πρόκειται να τροποποιήσετε την νομοθεσία σας ώστε να επισημαίνετε η παρουσία γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στα τρόφιμα. Και το θέμα της χρήσης ορμονών είναι πολύ σημαντικό και για σας και για μας. Γιατί βέβαια έχει απαγορευτεί η... Είναι λογικό να, να απαγορεύεται η εισαγωγή ε, κρέατος που έχει εκτραφεί με ορμόνες, γιατί απαγορεύεται αυτό από την νομοθεσία μας και παρόλα αυτά υπάρχει ένα τμήμα εισαγωγών που γίνεται. Μπορείτε να μας υποσχεθείτε ότι θα προσπαθήσετε να σεβαστείτε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όχι να προσπαθήσετε να την τροποποιήσετε. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ε, thank you very much. Ε, Ευχαριστώ. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τα όσα είπατε. Αναφερθήκατε ιδίως μεταξύ άλλων το καθαρισμένο με χλώριο σφάγιο είναι το αντίστοιχο με αυτό που δεν είναι. Γιατί η ορολογία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είπατε ότι αναθέσατε σε άλλους την ευθύνη να τρέχουν τις οικογένειές μας. Αν περάσει η TTIP όμως, θα, δώσουμε, θα αναθέσουμε την, το διατροφή των οικογενειών μας σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, ομίλους υπερκαταστημάτων. Μιλάτε τέλος για επιλογή των καταναλωτών. Αν ο καταναλωτής εκλέγει σε μια περιοχή τοπικές κοινότητες που δεν θέλουν γενελογικά τροποποιημένους οργανισμούς. Εμείς έχουμε πληροφορίες ότι το 2005 εσείς ψηφίσατε υπέρ ε, της απαγόρευσης στους, στις τοπικές κοινότητες να απαγορεύουν με τη σειρά τους την χρήση ε, γενεολογικά οργανισμών. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Υπουργέ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε μαζί σας. Πρώτα ερώτηση, μετά σχόλιο. Ακούσατε μάλλον για πολλές κόκκινες γραμμές. Ποιες είναι οι δικές σας κόκκινες γραμμές, σας ρωτήσω έτσι. Ποια είναι δηλαδή για σας τα παράβατα όρια. Και το σχόλιο τώρα στη δική μας περιφέρεια ένας από εμά πήγε σε μια αμερικανική περιοχή και καταστάθηκε Iowa Falls είναι στη δική σας πολιτεία μάλιστα εκεί που πήγα και τον είδα διαπίστωσα δύο πράγματα αφενός την ρεαλιστική προσέγγιση των Αμερικανών γεωργών που είναι πραγματικοί επιχειρηματίες και δεύτερον εντυπωσιάστηκα από την οικονομική και πολιτική ισχύ του, των αγροτικών συνεταιρισμών της ε, πολιτείας Αϊόβα. Κάτι που μπορούν να λάβουν σαν παράδειγμα και οι δικοί μας. Ο κ. Σεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Υπουργέ. Διακόπτη γιατί φαίνεται να υπάρχει κάποια σύγχυση. Ποιος είναι λοιπόν, ε, ποιος έχει σειρά. Α, εγώ, ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Υπουργέ. Εδώ στην Ευρώπη έχουμε πολύ υψηλά πρότυπα προστασίας των ζώων. Είμαι βέβαιος ότι τα πρότυπα αυτά τις επόμενες δεκαετίες θα βελτιωθούν κι άλλο, διότι οι πολίτες της Ευρώπης ενδιαφέρονται όχι μόνο για την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων, αλλά ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τον τρόπο που παράγονται τα τρόφιμα αυτά όλο και περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν να έχουν στα πιάτα τους το κρέας ζώων που έχουν υποστεί βασανιστήρια. Αυτά βεβαίως επηρεάζουν και τις τιμές παραγωγών. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι γεωργοί θα έχουν στην περίπτωση αυτή ένα ε, ανταγωνιστικό μειονέκτημα απέναντι στους Αμερικανούς. Εν τέλει βεβαίως οι τιμές των φτηνών προϊόντων θα είναι αυτές που θα κατησχίσουν. Η ερώτησή μου λοιπόν, θεωρείτε ότι μπορείτε να δεχτείτε και να υιοθετήσετε τα υψηλά πρότυπα προστασίας των ζώων που ισχύουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον Αμερικανό Υπουργό που είχε την καλοσύνη να έρθει και να συμμετέχει σε ανταλλαγή απόψεων. Καταρχήν, για το TTIP δεν είναι μόνο μια διαπραγμάτευση μεταξύ ε, κρατών ή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το TTIP είναι μια εταιρική σχέση που θα πρέπει να βρίσκει σύμφωνη και την κοινή γνώμη. Κατά τη γνώμη, κατά τη γνώμη σας, ε, σε αυτό το στάδιο, τι θα ήταν ποια θα ήταν η μεγαλύτερη υποχώρηση που θα μπορούσε να κάνει η κοινή γνώμη και θα ήταν το πιο δύσκολο που θα μπορούσε να αποδεχθεί το κοινό από τη συμφωνία αυτή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε επίγνωση του κινδύνου που δημιουργεί μικροβιακή αντοχή και μας ανησυχεί η εκτεταμένη χρήση αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς θα αντιμετωπίσετε, πώς θα αποσοβήσετε αυτό το φόβο των Ευρωπαίων και πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό. Κυρία Ριμπέιρο, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ καλό σημάδι για την πορεία των διατλαντικών σχέσεων. Και μάλιστα οι Αζόρες βρίσκονται ακριβώς στη μέση μεταξύ αυτών των δύο όχθων του Ατλαντικού. Ε, υπάρχουν προβλήματα με τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις προστατευμένε ονομασίες προέλευσης. Και αν δεν βρούμε λύση αυτό, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εγκρίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το TTIP. Είπατε για τις γεωγραφικές ενδείξεις ότι θα πρέπει να θετηθεί μια παράλληλη δράση. Τι εννοείται με παράλληλη δράση, ποια θα είναι η ε, παρέμβαση των κρατών μελών. Ε, θέλετε, και διμερεί σχέσεις ε, παράλληλα με το TTIP ή εκτός του TTIP. Ή τι, ποια είναι, θα είναι η παρουσία η παρέμβαση του, FDA, του Food and Drug Administration. Επίσης, η Πορτογαλία ενδιαφέρεται κυρίως ε, για το κρασί Πόρτο και το κρασί Μαδέρα. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και αυτών των γεωγραφικών ενδείξεων. Ποια είναι η γνώμη σας. Ο κύριος Νταντάν. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις να σας θέσω. Βλέποντας τη νέα αγροτική σας πολιτική, βλέπουμε ότι με αποφασιστικότητα η χώρα σας διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες. Οπότε δημιουργείται η ερώτηση. Θεωρείτε ότι η συμφωνία του Μαρακές έχει πλέον ε, καταπέσει, έχει πλέον, είναι απεχειωμένη όσον αφορά το, στο, τον ΠΟΕ έχετε έναν πρόεδρο, θα έχετε σε ένα χρόνο έναν εκλεγμένο πρόεδρο και έναν ενεργεία πρόεδρο. Μπορείτε πλην τις προεδρικές εκλογές να καταλήξετε κάπου και συναρτήσει των αποτελεσμάτων. Αν δεν υπογραφεί συμφωνία, είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν οι όροι της διαπραγματεύσεις προς κάποια κατεύθυνση, ή τη μία ή την άλλη. Ο Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που έδειξε και προλαλήσατε η κυρία Πετήρ για παράδειγμα, για τους μεταλλαγμένους οργανισμούς, τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Γιατί εμείς σταδιακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζουμε τη θέση μας απέναντι στους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, γινόμαστε όλο και πιο περιοριστικοί και πιο επιφυλακτικοί. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ε, πιθανότητα απαγόρευσης ε, των γενετικών γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στα κράτη-μέλη. Ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν τελείω διαφορετική πολιτική για τα μεταλλαγμένα. Ερωτώ λοιπόν, πώς ε, θα λάβει υπόψη ή δεν θα λάβει υπόψη η αμερικανική πολιτική την όλο και πιο στεντόρια φωνή των επιστημόνων, ακόμη και των Αμερικανών, εις βάρος των μεταλλαγμένων συστατικών. Γιατί ακούγεται ότι δημιουργούνται σοβαρές απειλές και κίνδυνοι από την χρήση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, που θα δυσκολέψουν ε, κατά πολύ τις εμπορικές μας ε, διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Ευχαριστώ κύριο Σκαλινόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Όταν δημοσιευθούν οι νέες διατάξεις με βάση τις οποίες και η Πολωνία είναι στον κατάλογο των χωρών που μπορούν να εξαγάγουν προς τις Ηνωμένε Πολιτείες τα μήλα που μας ενδιαφέρουν. Ε, πότε λοιπόν θα γίνει η δημοσίευση αυτών των διατάξεων, γιατί είχαμε ακούσει ότι θα δημοσιευθούν οι νέες διατάξεις μέχρι το τέλος του έτους. Είναι ορθό κάτι τέτοιο. Και εγώ έχω μία ερώτηση. Ποια είναι η γνώμη σας ε, για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Τι γίνεται. Ε, ποια είναι η εξέλιξη της, ε, των γεωρικών γεών την τελευταία δεκαετία. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των προδιαγραφών με βάση τα επιστημονικά κριτήρια. Γιατί οι συμφωνίες αυτές και μεταξύ μας, αλλά και οι συμφωνίες που γίνονται παγκοσμίω, θα, λάβουν, θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις νέες επιστημονικές εξέλιξεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε αυτό το σκέλος των συμφωνιών του TTIP. Uh, Βεβαίως Βεβαίω μεγάλος αριθμός ερωτήσεων. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω και σε συντομία βέβαια. Πάντως έχετε θέσει πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πρώτη ερώτηση. Γιατί δεν θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα φυτογειονομικών ως ένα ενίο μπλοκ, ένα ενίο συνασπισμό. Υπάρχουν διάφορα θέματα εδώ. Για παράδειγμα, όταν μια ζωνόσος ε, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, την ε, ε, γρήπη των πουλερικών δηλαδή, ένας αριθμός μόνο πολιτιών επλήγει από αυτές. Αν αντιμετωπίσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ενιαίο σχηματισμό, τότε εάν έχει πρόβλημα μία χώρα μέλος σας, θα αντιμετωπίσουμε ολόκληρη την Ευρώπη σαν να έχει ολόκληρη το ίδιο πρόβλημα. Γι' αυτό περνούμε μέσα από τις διαδικασίες που έχουμε θεσπίσει, που είναι ομοιόμορφες, και το ίδιο κάνουμε τώρα και για το βόλιο κρέα, είτε προέρχεται από την Ιρλανδία, είτε από την Ολλανδία, είτε από τη Λιθουανία. Προχωρούν αυτέ στο άνοιγμα τη Αμερικανική αγορά βόλιο κρέατο. Είναι φτιαγμένοι έτσι ώστε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα, εφόσον προκύψει κάποια ζωονόσος, με ε, τρόπο εξειδικευμένο. Δεν θεωρούμε ότι, για παράδειγμα, η πολιτεία της Βιρτζίνια επειδή μπορεί να έχει αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα μια ζωονόσου στην παραγωγή τη που θέλει να εξαγάγει ε, να πληγεί και το άνταχο που είναι χίλια χιλιόμετρα μακριά. Άλλο θέμα τώρα για το αμερικανικό ε, βόλιο κρέας. Ας το πω ως εξής. Εμείς έχουμε ένα σχετικά με, τα συνολικές, με τις συνολικές ποσοστώσεις με την ιδέα ότι θα έχουμε, μια, θα έχουμε μια ευκαιρία να χρησιμοποιούμε τα TRQ για να αντιμετωπίζουμε τις ζημίες στην αγορά του βόλου κρέατος. Έχουμε επιτρέψει ωστόσο σε εισαγωγές από ορισμένες άλλες χώρες να ε, εκμεταλλεύονται κάποια κενά στην νομοθεσία αυτή και να μπορούν να ε, εισάγουν περισσότερα στη δική μας αγορά. Ωστόσο πρέπει να υπακούσουμε στο πνεύμα του, της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και μετά από εκεί πέρα θα δούμε. Με ρωτήσατε επίσης σχετικά με το κόστος των προγραμμάτων που προέρχονται, που απορρέουν δηλαδή από τον Αμερικανικό νόμο Farm Bill. Κανένας από εμά δεν θεώρησε ότι πρέπει να πληρώνουμε τους γεωργούς ακόμα και όταν οι τιμές προϊόντων έχουν φτάσει σε ύψη ρεκόρ, ενώ αυτό γινόταν παλαιότερα. Ακόμα και όταν οι τιμές του καλαμποκιού ήταν πολύ υψηλές, λάμβαναν ενισχύσεις από την ε, κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Χρειάστηκε λοιπόν μεταρρύθμιση στην αγροτική νομοθεσία και θέλαμε ε, να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα προσφέρει ενισχύσει όταν αυτές πραγματικά απαιτούνται. 23 δισεκατομμύρια περίπου εξοικονομήσεις υπέρ του συνολικού προϋπολογισμού όταν πέρασε το ε, αγροτικό νομοθέτημα, το ΦΑΜΠΙΛ. Δεν είδαμε ε, απαραίτητα μεγάλη αύξηση των κονδυλίων για τον προϋπολογισμό για την έρευνα. Ωστόσο, για ορισμένα ιδρύματα ναι, τα οποία λάμβαναν 200 εκατομμύρια ε, δολάρια ίδρυμα ερευνών δηλαδή, λαμβάνουν και 200 εκατομμύρια από ε, ιδιωτικές επενδύσεις για την διεξαγωγή ερευνών στον αγροτικό τομέα, που ιστορικά είναι υποχρηματοδοτούμενες οι ερευνές αυτές εν ώψη και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε ε, τους όσους λαμβάνουν ε, πολιτικές αποφάσεις για να ενθαρρύνουμε τη σειρά τους την έρευνα, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα ε, ζωονόσους, ε, φυτογενομικά, ε, αλλαγή κλίματος, μέγα πρόβλημα το νερό, το οποίο πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος και εκεί χρειάζεται πολύς χρόνος και μεγάλη ε, προσοχή να του δοθεί σε όλες τις χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ελπίζω λοιπόν ε, να αυξηθούν οι υπολογισμοί για τα Ιδρύματα Ερευνών. με εντυπωσίασε ένα σχόλιο που άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με την ανάπτυξη με τρόπο που όχι η Αμερική, η Αμερική δηλαδή για την ανάπτυξη της υπέτρου. Εγώ μεγάλωσα ε, σε μια μεγάλη πόλη στο Πίτσπουργκ της Πενσιλβανίας. Με υιοθέτησαν και θα μπορούσα να πω ότι με ξαναϊοθέτησε η γυναίκα μου όταν παντρευτήκαμε και πήγαμε στο Άινταχο. Ε, εκπροσωπούσα τους γεωργούς ήδη από το 1980 όταν έγινε και μια σε βάθος μεταρρύθμιση της αγροτικής οικονομίας και πολλοί αγρότες τότε είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες και εγώ τους εκπροσωπούσα τότε. Εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ διότι έμαθα να αναγνωρίζω και να εκτιμώ οι άνθρωποι που δουλεύουν τη γη πόσο στενά συνδεμένοι είναι μαζί της. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω ό,τι μπορώ για να βελτιώσω τις οικονομικές τους δυνατότητες η πρόκληση που αντιμετωπίζαμε ήταν καθώς η αγροτική παραγωγή γινόταν πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική. Φτάσαμε από μια εποχή όπου 90% των Αμερικανών ήταν αγροτική οικονομία σε ένα 15%. Έχουμε τώρα τέσσερα θεμέλια παραγωγή, αγροτική παραγωγή. Εξακολουθεί να είναι σημαντική. Τοπικά συστήματα παραγωγή τροφίμων, που είναι που, πολύ, πολύ, σημαντικά για μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντο, του εδάφου. Αποφυγή τη διάβρωση των εδαφών. Διατήρηση τη ποιότητα. Και νέα ευκαιρία τώρα για τις αγορές, για την ε, αποφυγή έκκλησης διοξιδίων του άνθρακος. Πράσινη υποδομή, πράσινες υποδομές, πάλι για την διατήρηση. Πάλι επίσης πηγή εισοδήματο για τους αγρότες. Το ίδιο και ευκαιρίες αναψυχής, αναψυχής στις αγροτικές περιοχές, στην Ήπεθρο. Επίσης η χρήση ε, λιμάτων, γεωργικών λιμάτων που δεν είναι μόνο ίνες και υγραδίματα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως υποκατάστατα για πετρελαϊκά προϊόντα. Πάλι εκεί ανοίγονται ευκαιρίες δημιουργία θέσεων απασχόλησης και με τη χρήση των λιμάτων και της γεωργικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας και ούτω καθεξής. Και μιλούμε για μια αγορά της τάξης των 360 δισεκατομμυρίων τον χρόνο. Αρχίζουμε να βλέπουμε την γένεση μιας νέας οικονομίας bio-based που προσφέρει ε, έσοδα στους γεωργούς, δουλειές για όσους θέλουν να μείνουν στην Ήπεθρο και να αναθρέψουν τις οικογένειές τους. Υπάρχει λοιπόν και έχει και το Υπουργείο μου ένα σημαντικό συντελεστή ανάπτυξη της Υπέθρου, γιατί όπως σας εξήγησα ενδιαφέρομαι για τους ανθρώπους που ζουν στις μικρές πόλεις. Η γυναίκα μου από εκεί προέρχεται, έχω φίλους εκεί, τα παιδιά μου μεγάλωσαν σε μια μικρή πόλη και εκεί είναι και οι ψηφοφόροι μου που με εξέλεξαν εν τέλει βουλευτή και γερουσιαστή και θέλω να του εξασφαλίσω οικονομικέ δυνατότητε. Πολλέ ερωτήσει μου κάνατε για την επισήμανση, labeling δηλαδή. Έχουμε τώρα μια επισήμανση non-GMO, δηλαδή ότι δεν περιέχονται ε, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Όποιο θέλει να επισημάνει τα προϊόντα του ως non-GMO πρέπει να περάσει μέσα από μια διαδικασία για να επαληθεύσει ότι η επισήμανση αυτή είναι ορθή. Έχουμε και την βιολογική επισήμανση και συζητούμε τώρα στο Αμερικανικό Κογκρέσο την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένας κώδικας με γραμμές, ένας barcode δηλαδή και ενδιαφέρονται και μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή να διαθέτουν πληροφορίες τις οποίες μπορεί να σκανάρει κανείς με το κινητό του τηλέφωνο και να έχει αμέσως πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, εάν δηλαδή αυτό περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή όχι. Εάν όλα πάνε καλά, μπορούμε να δεχτούμε ένα σύστημα μηδενικής ανοχής. Με ρωτήσατε, όσο γίνονται οι μηχανισμοί ελέγχου πιο ακριβείς, θα είναι δύσκολο βέβαια να επιτευχθεί η τελειότητα, θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα να βάλουμε κάποιο κατόφλι να καθιδευτεί κάποιο κατόφλι αλλά νομίζω ότι μέσα στο χρόνο θα δείτε ότι οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν εάν κάτι που αγοράζουν είναι βιολογικό, είναι κάτι που δεν είναι βιολογικό αλλά δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή περιέχει και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και θα μπορούν να καταναλώνουν αντιστοίχως. Με ρωτήσατε αν έχω κόκκινες γραμμές. κόκκινες γραμμές έχει ο διαπραγματευτής για τη συμφωνία και μπορεί να μην χαρεί αν σας πω εγώ ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Δεν νομίζω ότι έχουμε καν κόκκινες γραμμές για την ώρα. Γνωρίζω ότι υπάρχουν δυσεπίλητα θέματα. Εσείς μάλιστα έχετε εντοπίσει ορισμένα όπως οι ε, γεωγραφικές ενδείξεις. Δύσκολο θέμα. Γιατί είναι δύσκολο. Έχουμε αγρότες στην Αϊόβα για παράδειγμα, στο Wisconsin, Καλιφόρνια που παράγουν τυρί που θεωρούν οι ίδιοι ότι θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τους γενώσιμους τίτλους για, για παράδειγμα ε, παρμεζάνα ή άλλα σχετικά να τα χρησιμοποιούν τα ονόματα αυτά αφού τα χρησιμοποιούν εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ο κόσμος εδώ στην Ευρώπη θεωρεί ότι θα πρέπει οι ονομασίες αυτές να χρησιμοποιούνται μοναχά από αυτούς που έχουν ξεκινήσει παραδοσιακά και τα χρησιμοποιούν. Εδώ παίρνουν δύο θέματα. Πρώτα, υπάρχει κάποια διαδικασία καθορισμού για, το, για, για την επαλήθευση, δηλαδή πραγματικά αυτό το προϊόν πράγματι ε, παρήχθη στο συγκεκριμένο μέρος που φέρει την ονομασία θήκε. Δεύτερο, πρέπει να κριθεί και το θέμα εάν η ονομασία έχει χρησιμοποιηθεί τόσο ευρέως και για τόσο πολύ μεγάλο χρόνο που τελικά να αποτελεί περιορισμό αυτών που παράγουν εάν τους απαγορευτεί να το χρησιμοποιούν. Εάν η γεωγραφική περιοχή παράγει το προϊόν θέλει να ε, χαρακτηρίζει το προϊόν, ίσως πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος, χωρίς να απαγορεύει την χρήση της γενώσιμης ονομασίας από άλλους. Στη συμφωνία TPP με την άλλη πλευρά του ειρηνικού δηλαδή, συζητούμε τις γεωγραφικές ενδείξεις και συζητούμε αυτές τις δύο προσεγγίσεις. Νομίζω ότι σε αυτές τις ε, δύο ε, προσεγγίσεις μπορούμε να βασιστούμε και για μια συζήτηση, για μια διαπραγμάτευση στην TTIP. Έχω βέβαια εδώ σελίδα ολόκληρη με τις ερωτήσεις σας, άρα μπορεί να μην τις απαντήσω με διαδοχική σειρά. Για τις εκλογές με ρωτήσατε. Βεβαίως και παίζουν σημαντικό ρόλο μπορεί ο νέος πρόεδρος να έχει διαφορετικές απόψεις ή να έχει και τις ίδιες απόψεις. Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι υποψήφοι για το προεδρικό αξίωμα που πιθανότατα θα λάβουν το χρήσμα των κομμάτων τους και κάποια στιγμή από αυτούς θα εκλεγεί και ο επόμενος πρόεδρος. Οι περισσότεροι από αυτούς λοιπόν υποστηρίζουν το ελεύθερο εμπόριο. Ίσως ορίζουν με διαφορετικό τρόπο το ελεύθερο εμπόριο, ίσως τονίζουν κάποιες άλλες πτυχές, ο ένας από τον άλλο δηλαδή. Οι περισσότεροι όμως, τουλάχιστον οι πιο σημαντικοί υποψήφοι για το προεδρικό αξίωμα, υποστηρίζουν γενικά τις εμπορικές ε, συναλλαγές. Υπάρχουν στοιχεία και στις ΗΠΑ όπως και στην Ευρώπη που έχουν πολύ έντονα συναισθήματα σχετικά με αυτά. Και στο δικό μου το κόμμα υπάρχουν ε, άνθρωποι και που εκπροσωπούν εργαζόμενους και ορισμένοι που εκπροσωπούν ε, αγρότες που έχουν εκφράσει αμφιβολίες και επιφυλάξεις για τις εμπορικές συμφωνίες. Από την άλλη ε, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις προϊόντων, εμπορικών προϊόντων, αγροτικών προϊόντων υποστηρίζουν τη συμφωνία αυτή. Βεβαίω είναι σημαντική η συζήτηση αυτή. Μέρο τη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ είναι ότι όσοι τάσσονται υπέρ της ελευθερία του εμπορίου δεν έχουν εξηγήσει καλά τα επιχειρήματά του και τη μεγάλη σημασία που έχει το εμπόριο για τη χώρα μας. Είναι εύκολο στη χώρα μου να κλείσει μια επιχείρηση και να ξανανοίξει, να ανοίξει στις ΗΠΑ και να ξανανοίξει κάπου αλλού και ο κόσμος θα ρίξει το φταίξιμο στο ελεύθερο εμπόριο. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι με, από την άλλη μεριά κάποιες μικρές επιχειρήσεις ανοίγουν θέσεις εργασίας, προσλαμβάνουν προσωπικό ακριβώς χάρη στην ελευθερία του εμπορίου. Αυτό όμως δεν φτάνει ποτέ στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νομίζω λοιπόν ότι οι υπέρμαχοι του ελεύθερου εμπορίου δεν έχουν προβάλλει με σωστό τρόπο τα επιχειρήματά τους. Ενώ οι άλλοι που έχουν ε, τις επιφυλάξεις το πράττουν με πολύ καλύτερο τρόπο. Θα δούμε βέβαια τους επόμενους μήνες με ποιο τρόπο θα ενημερωθούν ε, οι Αμερικανοί για τη σημασία του εμπορίου. Με ρωτήσατε και για μήλα και χλάδια. Ο κανόνας πάνω στον οποίο εργαζόμαστε στο Υπουργείο μου και βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια της ε, νομοθετικής αυτής ρύθμισης θα τα συζητήσουμε και με, αυτά, και με εσάς και θα τα έχουμε πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα αυτά. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, το θέμα αυτό είναι σημαντικότατο και πρόσφατα περάσαμε το νόμο για τον ξεχρονισμό της ασφαλείας των τροφίμων. Οι ΙΠΑ έχουν 15 οργανισμούς στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση που με κάποια μορφή είναι υπεύθυνε για την ασφάλεια των τροφίμων. Εγώ και ο πρόεδρο αναφέραμε ότι θα πρέπει να έχουμε έναν ενίο φορέα επιφορτισμένο από την ασφάλεια των τροφίμων. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε με την νομοσχέδιο εξυγχρονισμό τη ασφάλεια των τροφίμων να παραλληλήσουμε με αυτό που γίνεται από το, από το Υπουργείο Γεωργία, από την, ε, την Οργανισμό για τα Τρόφιμα που ελέγχει 80% των τροφίμων. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει τα επεξεργασμένα αυγά, ε, τα πουλερικά και το κρέας. Αν παραγγείλει μία πίτσα στι ΗΠΑ, ποιο είναι το παράδοξο. Και έχει απλώς τυρί πάνω τη. Θα ρυθμίζει ε, η υπηρεσία τροφίμων. Αν βάλετε και ένα σαλάμι πάνω, ένα κομμάτι σαλαμιού, τότε το Υπουργείο Γεωργίας είναι υπεύθυνο. Αυτό δεν έχει δεν, νόημα. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Καταρχάς να ευθυγραμμίσουμε τα προγράμματα, διότι η FDA, ο Οργανισμό Τροφίμων, ανταποκρίνεται σε πρόβλημα κυρίως. Ενώ το Υπουργείο Γεωργίας αντιδρά όσον αφορά την πρόληψη. Πώς ξεκινάς από το να προλάβεις το πρόβλημα. Οπότε έχουμε πολύ αυστηρούς ελέγχους και πρόσφατα μεταρρυθμίσαμε και το όλο σύστημα ελέγχων και επεκτείναμε ε, και τα, διάφο τα διάφορες ουσίες που ψάχνουμε να βρούμε και αν υπάρχει πρόβλημα στο τρόφιμο τελικά ε, τα απαγορεύουμε. Λοιπόν, Θέλουμε καλύτερη ευθυγράμμιση όσον αφορά τα συστήματα για την ασφάλεια των τροφίμων και σε κάποια φάση να είναι ευκολότερο αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ενιαίο φορέα για την ασφάλεια των τροφίμων, να είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτή η κίνηση. Προφανώς είναι σημαντικό να υπάρχει έλεγχος απονομή ευθυνών, απόδοση ευθυνών και θα πρέπει να αντιδρούμε αν υπάρξει πρόβλημα την ασφάλεια των τροφίμων, να υπάρχει χνηλασιμότητα, και με 300 εκατομμύρια καταναλωτές και πάνω από ένα τρισεκατομμύρια πιθανότητε να μηνθεί πρόβλημα το χρόνο, όλα αυτά τα θέματα ασφαλεία των τροφίμων είναι κάτι ε, πάρα πολύ σοβαρό. Όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την ευημερία των ζώων, ε, εμεί ε, τη βιωσιμότητα γνωρίζουμε ω εξή. Λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο την κοινωνική βιωσιμότητα, Εκεί εμπίπτουν και οι κανόνε στην ευημερία των ζώων, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα λαμβάνονται υπόψη. Και αν θέλουμε να έχουμε σύστημα βιώσιμο ή βιωσιμότητα, δεν μπορεί να έχει ένα ή δύο. Πρέπει να καλύπτει και τι τρει στοιχείε. Μπορεί να έχει υψηλότερε προδιαγραφέ, πολύ ψηλέ προδιαγραφέ, αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστούν, δεν θα εφαρμοστούν. Μπορεί να έχει τι πιο φθηνέ προδιαγραφέ, οπότε εκεί θα έχει προβλήματα όσον αφορά την ευημερία των ζώων και ίσω το περιβάλλον. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπου με του οποίου να έχουμε βιωσιμότητα συνολικά και όσον αφορά την ευημερία των ζώων, ε, συνεργαζόμαστε με αρμόδιου φορεί για να δημιουργήσουμε προδιαγραφέ, ούτω ώστε να υπάρχουν σαφεί κανόνε προαπαιτούμενα, να επικρατεί διαφάνεια όσον αφορά τι προδιαγραφέ. Και θα γίνουν τα δέοντα και η αγορά παίζει σημαντικότατο ρόλο. Οι καταναλωτές είναι απαιτητικοί και η αγορά ανταποκρίνεται. Κάποια από τα μεγαλύτερα εστιατόρια fast food αλλάζουν την προσέγγιση τους διότι τα πετούν οι καταναλωτές και θα δείτε να γίνεται όλο και περισσότερο αυτό στο μέλλον. Έγινε κάποια κουβέντα μεταξύ ταυτοσύμωσης συστημάτων και ισοδυνάμων και μετέθεσαν ερωτήσεις. Να πω ειλικρινά ότι αυτό απαιτεί επίπεδο συζητήσεως που δεν μας επιτρέπει σήμερα ο χρόνος. Ε, αλλά να πω τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να πω το εξή. Μέσω παραδείγματα, στα βιοκαύσιμα Φερρυπίν. Εσείς υποστηρίζετε τα βιοκαύσιμα, την έννοια των βιοκαυσίμων, αλλά μόνο αν ε, ήταν παράγονται με βιώσιμο τρόπο οι ζωοτροφές. Αυτοί παράγουν σόγια, πιστεύουν οι γεωργοί μας ότι παράγουν βιώσιμα τη σόγια. Όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως στην Ευρώπη, αλλά νομίζουν ότι περιμένουν το ίδιο τελικό αποτέλεσμα μέσω της δικής του διαδικασίας. Για μας αυτή είναι μια ισοδυναμία, αλλά δεν είναι ταυτόσιμα τα συστήματα. Είναι ισοδύναμα. Αν καθορίσετε τον στόχο σας, τότε το ερώτημα είναι μόνο με έναν τρόπο πετυχαίνει το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλαπλή τρόποι για τον ίδιο στόχο. Αν υπάρχουν πολλαπλή τρόποι μπορεί να έχετε ισοδύναμα συστήματα που δεν είναι απαραίτητα τα ίδια. Αυτές οι συζητήσει θα εκτελεχθούν στο TTIP, θα γίνει πολλή κουβέντα γι' αυτό. Τι προσπαθούμε να πετύχουμε, ποιο είναι το ευθέο αποτέλεσμα, μόνο με έναν τρόπο το πετυχαίνουμε. Το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων ήταν κάτι σημαντικό που συζητήσαμε. Γεωγραφική ένδειξη προέλευσης, γεωγραφική ένδειξη είναι ε, ο μόνος τρόπος ή και το εμπορικό σήμα είναι ένα άλλο τρόπος. Ή να συνδυάσουμε τα δύο που ίσως ε, τελικά μπορούν να οδηγήσουν σε λύση. Α, ρωτήσατε για την ερώτηση της μικρής εκμετάλλευσης, για το θέμα, τον ορισμό της μικρής εκμετάλλευσης. Έχουμε 2,2 εκατομμύρια αγρότες στις ΗΠΑ, όπως τους καθορίζουμε εμείς σαν γεωργούς. Γεωργός είναι εκείνος που παράγει προϊόν, σύμφωνα τον ορισμό μας, το οποίο προϊόν έχει μία αξία ε, χιλίων δολαρίων και πάνω στην πώληση. Είναι ευρύ ορισμό του γεωργού. Αλλά εντό των 2,2 εκατομμυρίων γεωργών έχετε περίπου 1,3 εκατομμύρια γεωργού οι οποίοι παράγουν προϊόντα που ίσω να, ανήκουν, να έχουν μια αξία λιγότερη από 10.000 δολάρια. Η τεράστια πλειοψηφία εκείνων που ορίζουμε ω Γεωργιού, η πλειοψηφία από αυτού, είναι σε αυτή την κατηγορία. Παράγουν λιγότερα από 10.000 ίσως κάτι να φτιάχνουν στο σπίτι τους, να το πουλούν οι στην αγορά, στην τόπια αγορά να πηγαίνουν και να παράγουν ε, κρασί από μήλο, μιλίτη και υπάρχουν λίγοι που παράγουν κάτι παραπάνω από 10.000 και λιγότερο από 250.000, μικρό ποσοστό. Αυτούς τις είπα θα τους έλεγαν σαν οικογενειακές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκείνη είναι εκείνη που θα ορίζατε στις ίπα σαν οικογενειακές επιχειρήσεις, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Οπότε μας μένουν περίπου 200.000, 200 με 300.000 παραγωγοί που παράγουν πάνω από 250.000 δολάρια ε, είναι η παραγωγή μεγάλης κλίμακας. εκμεταλλεύσουμε μεγάλη κλίμακας παράγουν σημαντικό ποσοστό των παραγωμένων στη ΣΥΠΑ, όσον αφορά τους αριθμούς ανθρώπων είναι σχετικά λίγοι. Η τεράστια πλειοψηφία των γεωργών είναι στην κατηγορία των μεσαίων μικρομεσαίων και πολλούν λιγότερα σε ποσά κάτω των 25.000 δολαρίων και σε αυτού που είναι κάτω από 10.000 και σε αυτού που είναι κάτω από 250.000 όλοι αυτοί είτε οι ίδιοι είτε οι σύζυγοί του πρέπει να εργάζονται στην εκμετάλλευση. Γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε μια παράλληλη συνοδευτική οικονομία να του δίνει δυνατότητε και νέες πηγές εισοδήματος ώστε να του διευκολύνουμε, να μπορούν να κρατήσουν την εκμετάλλευση χωρί να πρέπει να έχουν δύο δουλειέ. Διότι αντιμετωπίζουμε την εξή κατάσταση. Οι νέοι που βλέπουν πόσο σκληρά εργάζονται οι γονεί του, δεν θέλουν να ασχοληθούν απαραίτητα με τον Γεωργέτσο, αρέσει τόσο το τελευταίο που θα είχα να πω τώρα. Αφορά ε, βιολογικά και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, βιολογικά προϊόντα παράλληλα, αυτά τα δύο. Πριν από δύο χρόνια ξεκίνησε η συζήτηση. Το NC21 το ονομάσαμε το πρόγραμμα. Έχουμε 21 ανθρώπους εκεί που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα ε, της, της γεωργίας παράγουν βιολογικά προϊόντα, γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, ε, ανήκουν σε ομάδες προβληματισμούς για τη γεωργία και τους είπα, σκεφτείτε πώς η βιολογική παραγωγή, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, όλοι αυτοί, όλες οι παραγωγές μπορούν να συνεπάρξουν και έκανα κάποιες συστάσεις. Ε, μία φορά τον έλεγχο, την ανάγκη παραγωγή να καταλάβουν τι κάνουν οι γείτονές τους, να υπάρχει κάποια συλλογική προσέγγιση και αυτοί που παράγουν σπόρους, οι εταιρείε να γνωρίζουν πότε είναι σωστός χρόνος, σωστή μέθοδος και σωστός τόπος για να φυτευτούν οι σπόροι, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους για να μειωθούν οι κίνδυνοι. Μετά υπήρχε και η ανάγκη για πρόσθετα εργαλεία για τη διαχείριση του κινδύνου για βιολογικούς παραγωγούς και το πώς θα ασφαλίζονται οι βιολογικοί παραγωγοί, το αλλάξαμε αυτό την ασφάλιση και πώς καταβάλλεται αποζημίωση περίπτωση προβλήματο. Τρίτον, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τη δυνατότητα επιμόλυνσης από γειτονικέ ε, καλλιέργειες. Ανακαλύψαμε πράγματα όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεν είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα όσο νομίζαμε. Η επιμόλυνση από το τριφύλι παραδείγματο χάρη εξετάσαμε. Ε, δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα και κάναμε έναν έλεγχο σαν φάση βιολογικούς παραγωγού και ρωτήσαμε πόσοι πολλοί είχατε προβλήματα μόλυνσης και είναι πραγματικά, πραγματικά πολύ χαμηλό το ποσοστό. Η ερώτηση είναι πόση βιολογική παραγωγή υπάρχουν στην, ε, στη ΣΥΠΑ. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Περίπου 20.000 άνθρωποι επίσημα έχουν επιστοποιηθεί ότι είναι βιολογική παραγωγή. Πιθανότατα υπάρχουν και άλλοι που διαθέτουν τα προϊόντα στην αγορά, βιολογικά προϊόντα, που δεν πέρασαν ε, τη διαδικασία επιστοποίηση, αλλά μπόρεσαν να καλύψουν τι ανάγκε και να πληρούν τι προποθέσει. Επίσημο αριθμό είναι περίπου 20.000 αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να... Δεν ξέρω ποια ήταν αυτή η ψήφο το 2005. Ήμουν κυβερνήτη τότε. Δεν ήμουν στην νομοθεσία. Δεν ψήφισα. Δεν ξέρω περί τίνο πρόκειται. Αν θέλετε να μου δώσετε περισσότερε πληροφορίε, με τα χαρά να προσπαθήσω να σα δώσω κάποιε εξηγήσει, να σα εξηγήσω περί τίνο πρόκειτο. Κοιτάξτε, οι εφημερίδε από ό,τι ξέρω δεν τα λένε πάντα σωστά δεν έχουν πάντα δίκιο, ίσως να αληθεύει αυτό που λέτε, ε, νομίζω ότι κάλυψα τις περισσότερες ε, ερωτήσεις, ίσως κάποιες να μου ξέφυγαν, αλλά ήταν καλή η συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Πληθώρα ερωτήσεων, ε, πολύ διαφορετικό μεταξύ τους μάλιστα. Βλέπετε από το χειροκρότημα πώς εκτιμούμε την παρουσίαση εδώ και την ανταλλαγή απόψεων. Ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπατε στην αρχή. Είπατε ότι η γεωργία δεν γίνεται κατανοητή πάντα στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, σημαντικό το μήνυμα γιατί αυτή την αίσθηση έχουμε και εμείς, ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει επαρκώς τη γεωργία και τη σταπή γεωργία και τη συνεισφέρει γεωργία. Γιατί είναι πολύ σημαντική η συμβολή της και έχει σχέση και με άλλους τομείς. Σε ό,τι αφορά την επιθετιστική ασφάλεια, κατά τη γνώμη μου ε, θα πρέπει το TTIP να ενισχύει αυτή την ε, επιστηστική ασφάλεια συμβάλλοντας σε μια κοινή αντίληψη για την γεωργία. Γιατί από τη στιγμή που είμαστε σε παγκοσμιοποιημένο κόσμο θα πρέπει να έχουμε κοινή αντίληψη και για τη γεωργία, όπως συμβαίνει και για τα χρηματοπιστωτικά θέματα. Και η γεωργία επίσης χρειάζεται παρεμβάσεις μερικές φορές. Γιατί από μόνη της δεν τα καταφέρνει πολλές φορές. φαίνεται ότι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος είναι πιο αυτόνομος και τα καταφέρνει καλύτερα και χωρίς παρέμβαση από τη Γεωργία. Η Γεωργία όμω επηρεάζεται και από εξωτερικούς παράγοντε πολλούς, Γι' αυτό και χρειάζεται βοήθεια μερικέ φορέ. Επηρεάζεται από τι κλιματικέ αλλαγέ, για παράδειγμα. Επίσης, μιλήσετε για την δημογραφική αύξηση. Το 2050 θα είμαστε 7 δισεκατομμύρια. Θα αυξηθούν οι επιστημιστικές ανάγκες σε συγκεκριμένες χώρες επίσης, αλλά θα έχουμε πρόβλημα και με το νερό, με τη λειψιδρία, το θέμα το, της υφαρπαγής των γεών, το land grabbing, έχουμε απώλεια γεωργικών εδαφών. Πολύ σημαντικές αυτές οι προκλήσεις και επιβαρύνουν τη γεωργία και τους γεωργούς. Γι' αυτό και όπως είπα ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων και ελπίζουμε για πολλά θέματα να έχουμε σύγκληση. Αλλά μετά από αυτά που είπατε, αυτή την αίσθηση είχαμε ότι υπάρχουν αρκετά σημεία σύγκληση. Αν και εγώ πιστεύω ότι οι διαφορές είναι παρόλα αυτά βαθιές. Γιατί ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε μια νέα γεωργία. Άλλα χαρακτηριστικά έχει η γεωργία του Βόρα και άλλα η γεωργία του Νότου. Και νομίζω ότι οι εσωτερικέ μα διαφορέ είναι πολύ μεγαλύτερε από ό,τι οι εσωτερικέ διαφορέ τη γεωργία στι ΗΠΑ. Μα περιπτώσει, θερμά ευχαριστώ για τη συμμετοχή σα. Σίγουρα θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Αλλά όπω είπα, η ανταλλαγή απόψεων ήταν πολύ χρήσιμη για μα. Σα ευχαριστούμε θερμά. Ε, πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω ξανά για τη δυνατότητα που μου δώσατε και εκτιμώ το χρόνο και την προσοχή που μου δώσατε. Δύο πράγματα να πω, κλείνοντας. Πρώτα απ' όλα, η Ευρώπη έχει μεγάλη, πολύ καλή φήμη. Οι Ευρωπαίοι γεωργοί, τα ευρωπαϊκά προϊόντα έχουν άριστη φήμη. Είναι προϊόντα με ύψιστη προστιθέμενη αξία. Είναι προϊόντα που οι Αμερικανοί ε, καταναλωτές ε, τα εκτιμούν και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ενισορροπία μεταξύ ΙΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα προϊόντα, διότι είναι πολύ ψηλή η ποιότητα των προϊόντων. Και είπατε σε μια ερώτηση πώς μπορεί να επιβιώσει την όλη δικασία Ευρώπη. Επιβιώνει συνεχίζοντας να εστιάζεται επί προϊόντων της ποιότητας. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, εμείς συλλογικά όσοι ενδιαφερόμαστε για τη γεωργία έχουμε δύο σημαντικά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα θα αντιμετωπίσουμε σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά το κλίμα. Και σαν τομέα σαν λαοί, σαν, σφαιρικός, σαν παγκόσμιος πρέπει να κινηθούμε σοβαρά. Και θα πρέπει να εστιαστούμε από αυτού στο Παρίσι. Και δεύτερον, σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες εγώ πάντα ανησυχούσα για το θέμα το πώς μπαίνουμε όσον αφορά την οικονομία. η αριθμή των γεωργών στη ΣΥΠΑ είναι πολύ μικρός. Και δεν συζητούμε τόσο πολύ τους ελέγχους, δεν έχει τέτοια προτεραιότητα. Ίσως φαρμακευτικά, αυτοκινητοβιομηχανία κλπ. να έχουν μεγαλύτερη σημασία. Σειρά άλλων θεμάτων που είναι πραγματικά πολύ σημαντική παράγοντα στην οικονομία. Αλλά αυτό που ακούστηκε πριν είναι το εξή. Αν δεν υποστηρίξουμε του γεωργού και τελικά χρεοκοπήσουν και δεν εργάζονται πλέον οι γεωργοί, δεν έχει καμία σημασία τι θα συμφωνήσουμε όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Θα πρέπει η γεωργία, οι ηγέτες δηλαδή, σε όλες τι χώρε που διαμαγωτεύονται τη γεωργία, να εκτιμήσουν το σημαντικό ρόλο των γεωργών και να θα πρέπει να τους σέβονται και εγώ το λέω κυρίω για τους δικούς μου, το δικό μου λαό, να εκτιμούν τους γιοργού, να εκτιμούν αυτό που κάνουν. Διότι τους αναθέσαμε πολύ σοβαρή ευθύνη. Δώσαμε πολύ σοβαρή ευθύνη σε πολύ λίγους ανθρώπους, μας δώσαν την ελευθερία εμείς να επιδιώξουμε, πετύχουμε τα όνειρά μα και δεν του έχουμε ευχαριστήσει ποτέ αρκετά γι' αυτό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε και πάλι θερμά κύριε Υπουργέ. Κατά τη γνώμη ήταν πολύ χρήσιμη και πολύ επικοδομητική αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Και σίγουρα θα επανέλθουμε σε αυτό που μας είπατε αρκετές φορές. Μία ολιγόλεπτη διακοπή για να ξεπροβοδίσουμε τον κύριο Υπουργό.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 Έχουμε μείνει λίγο πίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, γι' αυτό περάσουμε γρήγορα στο σημείο 5 της τη διάταξης. Δεν ξέρω ποια σειρά θα ήταν η καταλληλότερη, ποιο σημείο θα έπρεπε να προηγείται και ποιο να έπεται. Εν πάση περιπτώσει πάμε στο σημείο 5, ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, διαπραγματεύσεις στο θέμα της γεωργίας στο πλαίσιο του TTIP. Έχουμε τον αρμόδιο επικεφαλής ε, διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γεωργία στο TTIP, τον ε, ασκώντα καθήκοντα Γενικού Διευθυντού στη Γενική Διεύθυνση Άγκρη, τον κύριο Τζον Κλάκ, αναπλήρωτο του Γενικού Διευθυντού. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα Γι' αυτό θα ήθελα ερώτηση. Αναμεταδίδεται η συνεδρίασή μας είναι και κλεισμένα το θυρών, αυτό το τμήμα της τουλάχιστον. Ναι, ναι, μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Δεν είναι και κλεισμένο το θυρών. Θα σας δώσω το λόγο αμέσω, κύριε Κλάρκ. Λάβετε υπόψη παρακαλώ την ε, καθυστέρηση. Βέβαια δεν φταίτε εσείς, ούτε και σας αφορά το γεγονός ότι καθυστερήσαμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν κανείς ανεβαίνει στη σκηνή δεν θα πρέπει να συναγωνίζεται ούτε ζώα ούτε παιδιά. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι αδύνατο να συναγωνιστώ τον ε, προηγούμενο καλεσμένο, τον Τόμ Βίλσακ, τον ε, Υπουργό Γεωργίας Αμερικής. Ε, ήταν απαράμιλη δική μου ομιλία. Εγώ θα σας δώσω μια πιο ε, ταπεινή και μετριόφρονα ευρωπαϊκή προσέγγιση για το γεωργικό σκέλος του TTIP μετά τις διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των ε, ήδη συστομένων γεωργικών συμφωνιών, ε, εμπορικών συμφωνιών. Και τέλος αυτό που είπε στο τέλος ο κύριος Βίλσακ, ότι το θέμα της επιστημικής ασφάλειας και της διεθνούς συνεργασίας επίσης θα αναφερθεί. Τώρα κάποια πρακτικά στοιχεία. Συμφωνούμε ότι ε, η ΚΑΠ είναι σημαντικότημα του εμπορικού μας προγράμματος και των εμπορικών μας διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να αποδείξουμε στους φορολογουμένους μας ότι και τα γεωργικά προϊόντα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, όπως και η παραγωγή άλλων προϊόντων. Συμβάλλουμε λοιπόν με τη γεωργία στην αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη και οι εξαγωγές μας είναι 2,2 ε, στηρίζουν άμεσα 2,2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Και αν ρίξετε μια ματιά στον πίνακα που βλέπετε στις οθόνες σας, διαπιστώνετε ότι για τέταρτη συνέχεια χρονιά είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, ενώ παλιά ήμασταν εισαγωγής, ε, μεγαλύτερη εισαγωγής ε, γεωργικών προϊόντων. Πάνω από τη, μέση, τη γραμμή, τη μεσαία είμαστε στις εξαγωγές, κάτω είμαστε στις εισαγωγές. Βλέπετε υπάρχει αύξηση των εξαγωγών στο ισοζύγιο το γεωργικό. Και βάλιστα δεν εξάγουμε μόνο προϊόντα υψηλή προστιθέμενες αξίες, αλλά και ενδιάμεσα προϊόντα, αλλά και βασικά προϊόντα, όπως δημητριακά για παράδειγμα. Το 2015 η ίδια θετική τάση συνεχίζεται παρά το ρωσικό εμπάργο στο τέλη του 2014 που επηρέασε ε, εξαγωγέ μας ύψου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζουμε παρόλα αυτά την αύξηση των εξαγωγών και μάλιστα αναμένεται αύξηση γύρω στα 6% το χρόνο στις εξαγωγές μας. Οι μελλοντικέ προοπτικές είναι γενικώ θετικέ. Η αύξηση τη ζήτηση εντό Ευρώπη θα παραμείνει σχετικά χαμηλή, αλλά όπως είπε και ο Υπουργός Βίλσακ, υπάρχει τεράστια αύξηση της ζήτησης στις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας, αλλά και στις αφρικανικές χώρες. Από εκεί θα έχουμε και σημαντική δημογραφική αύξηση, μεγαλύτερη ε, μεσαία τάξη την επόμενη τριακονταετία και, και άρα αύξηση της ζήτησης ε, πρωτεϊνών, κρέατος, ε, με μεταποιημένων επεξεργασμένων προϊόντων και άρα θα αυξηθούν και οι δυνατότητες εξαγωγής τέτοιων προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε εδώ τα διάφορα μοντέλα εισαγωγών-εξαγωγών, περσινές εισαγωγές. Οι εισαγωγές μας ήταν κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία, βασικά προϊόντα, σόγια, ζωοτροφές, ξηρούς καρπούς, από την Κίνα κάποια απορροκυπευτικά, από την Ινδονησία φινικέλαιο. Κυρίως εισάγουμε βασικά προϊόντα που τα μεταποιούμε στη συνέχεια, περαιτέρω, και το ρεάλι όψη του νομίσματος, οι εξαγωγές δηλαδή, αυτές είναι οι μεγαλύτερες μας αγορές, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Νοτιοανατολική Ασία, Κίνα, Μέση Ανατολή, μεγάλη αγορά για τα δημητριακά μας και από μέχρι τα μέσα του περσινού χρόνου και η Ρωσική Ομοσπονδία ήταν σημαντική αγορά για τις εξαγωγές μας. Τώρα για το πρόγραμμα του ΠΟΕ. Δέκα μέρες μας χωρίζουν από την Υπουργική Διάσκεψη του Ναϊρόμπι και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η πρόσβαση στις γεωργικές αγορές και το θέμα των, ε, των επιχορηγήσεων δεν θα τεθεί στη ημερήσια διάταξη του Ναϊρόμπι. Μόνο ο ανταγωνισμός στις εξαγωγές ε, θα συζητηθεί και μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα ιδιαίτερος. Αυτό που θα επιδιώξουμε στη Υπουργική Διάσκεψη του Ναϊρόμπι είναι μια ισορροπία ώστε να μην επικεντρωθούμε μόνο στις ε, εξαγωγικές ε, επιδοτήσεις γιατί υπάρχει πρόταση για μόνιμη κατάργησή τους και αυτό θα καταστεί δυνατό να γίνει στο Ναϊρόμπι μόνο αν ταυτόχρονα και ε, ή εξαγωγικές πιστώσεις ή κάποιες μορφές επιστηστικής βοήθειας και άλλες μέθοδοι που παρομοιάζουν με αυτές των εξαγωγικών επιδοτήσεων και αυτές καταργηθούν. Δεν μπορούμε και εμείς μόνο μερός να καταργήσουμε τις εξαγωγικές μας επιστροφές όταν δεν γίνουν άλλες χειρονομίες από εταίρους μας. Τώρα, για τις διμερείς μας διαπραγματεύσεις. Εδώ και αρκετά χρόνια, μεγάλο τμήμα του εμπορικού μας θεματολογίου αφορούσε διμερείς εμπορικέ συμφωνίε και μάλιστα επειδή δεν είχαμε συμφωνία στον ΠΟΕ για τη γεωργία, ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε τους δασμούς στις αγορές μας για τις εξαγωγές ήταν μέσω διμερών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Και αυτός ο χάρτης δείχνει τι διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου συνήψαμε τα τελευταία δύο με τρία χρόνια. Είχαμε την Κορέα, την Κολομβία, τον Περού, τον Καναδά, την Νότια Αφρική, και τις τελευταίες εβδομάδες ε, συνήθως συμφωνία, ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις και με συμφωνία για το Βιετνάμ. Σημαντικό θέμα, γιατί το Βιετνάμ απελευθέρωσε πλήρως όλους τους τομείς που μας ενδιαφέρουν για τις εξαγωγές. Βόλιο, κρέας, χείριο, γαλακτοκομικά, ε, ίνος και ίνοπνευματόδη και ένα μεγάλο φάσμα γεωργικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές μας από το Βιετνάμ, Φροντίσαμε για τους ευαίσθητους τομείς μας, το ρύζι, το άμυλο και τη ζάχαρη, όχι μέσω πλήρους απελευθέρωσης, αλλά μέσω ποσοστώσεων δασμολογικών. Και μάλιστα μέσω της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου με το Βιετνάμ έχουμε πλήρη προστασία 170 σημαντικότερων προϊόντων μας που ε, χαίρουν γεωγραφικής ένδειξης. Έτσι θα έχουμε πρόσβαση σε μια αναπτυσσόμενη αγορά 9 εκατομμυρίων, 90 ε, ναι, συγγνώμη εκατομμυρίων, το Βιετνάμ, και ταυτόχρονα θα μας βοηθήσει στην περαιτέρω ε, επέκτασή μας στην εμπορική, στην νότιο και νοτιοανατολική, ανατολική και νοτιοανατολική Ασία. Ποια θα είναι η επόμενη φάση τώρα διμερών ε, συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Ε, για την Κίνα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει για τι γεωγραφικέ ενδείξει. Με χώρε του Περσικού κόλπου επίση και με την Ιαπωνία έχουμε διαπραγματεύσει. Η Ιαπωνία σημαντική αγορά για τα αγοραπιστιστικά. Είναι μια αγορά πολύ προστατευμένη και για τα γεωργικά προϊόντα και για τις γεωργικέ ενδείξεις. πάντω προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε πολύ φιλόδοξη έκβαση των διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία. Δεν θα μας αρκέσει μια χαμηλή φιλοδοξία σαν αυτή που χαρακτήρισε την ε, Συμφωνία του Ειρηνικού, την εταιρική σχέση του Ειρηνικού. Θέλουμε ένα υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας. Και δεν θέλουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση τους ε, εξαγωγείς μας με χαμηλές φιλοδοξίες. Μιλήσατε το απόγευμα για το TTIP. Αυτές είναι οι 10 μία από τις 10 προτεραιότητες της Επιτροπής και του προγράμματος Juncker. Στόχος μας είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των επιθετικών και των αμυντικών μας συμφερόντων. Γιατί έχουμε ε, εμπορικά συμφέροντα στην Αμερικανική αγορά, κυρίως για τα γαλακτοκομικά, κάποια προϊόντα κρέατος και για τον ίνο ε, το ενοπνευματώδη και την προστασία γεωγραφικής ένδειξης. Και έχουμε και κάποιες ευαισθησίες και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί γι' αυτό. Το επισήμανε εύστοχο ο κύριο Νίκολσον. Βόλιο, πουλερικά, χείριο, κρέα ρύζι σε κάποιο βαθμό, άμυλο, εθανόλη. Εκεί το κόστο παραγωγή στην Ευρώπη είναι υψηλότερο από ό,τι στι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε διαφορετικέ οικονομίε κλίμακο και άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο ανταγωνιστικέ στον τομέα αυτό. Οπότε σε μια συμφωνία εταιρική σχέση τύπου TTIP δεν θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε πλήρω του τομεί αυτού. Ε, στη δική μας αγορά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αλλά θα πρέπει να βρούμε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, ανοίγοντας κάποιες δοσμολογικές ποσοστώσεις, δίνοντας στις ΗΠΑ ε, κάποια βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά μας, χωρίς όμως να υπονομεύουμε τη θέση των γεωργών μας και της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Νομίζω ότι αυτό το αναγνώρισε ο Υπουργό Βίλσακ όταν είπε ότι πρέπει να μειωθούν. Ίσως να προστατεύσουμε τη, τη γεωργία ώστε να μην μειωθεί υπερβολικά ή να μην εξαφανιστεί ο γεωργικός ιστός. Τώρα, όπως σας είπα, μερικοί τομεί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, αλλά σίγουρα η κόκκινη μας γραμμή είναι τα φυτογενομικά μας πρότυπα και οι φυτογενομικές προδιαγραφές. Το επαναλαμβάνω, το ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπονομεύσει τα ε, υγειονομικά και φυτογειονομικά μας πρότυπα για τα τρόφιμα. Δηλαδή, όχι κρέας με ορμόνες, ούτε χλωριοποιημένα κοτόπουλα δεν θα φτάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή στα πιάτα μας. Είναι αδιαπραγμάτευτες αυτές οι προδιαγραφές. Μία σημαντική συμφωνία που θα ξεκινήσει μάλλον στο εγγύς μέλλον, αλλά με δυνητικό αντίκτυπο σοβαρό για την Ευρωπαϊκή Γεωργία, γι' αυτό θα πρέπει να γίνει σοβαρή αξιολόγηση, είναι με το Μερκοσούρ, που όπως οι ΗΠΑ είναι σημαντικός ανταγωνιστής ε, στο κρέας, ε, σε βασικά προϊόντα, στη ζάχαρη και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους τομείς αυτούς σε μια μελλοντική διαπραγμάτευση με το Μερκοσούρ. Ίσως διαβάσατε την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής για την στρατηγική στις επενδύσεις για το εμπόριο. Είναι αρκετά φιλόδοξο το πρόγραμμά μας εν ώψη και των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου. Θα ζητήσουμε εντολή από το Συμβούλιο ώστε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία καθώς και με το Μεξικό και τη Χιλή. Οπότε αν ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις θα προσθεθούν στις διαπραγματεύσεις που έχουμε με εξίσου ανταγωνιστικές χώρες όπως είναι το Μερκοσούρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό και ο αρμόδιος επίτροπος δεν χάνει την ευκαιρία να τονίσει την ανάγκη μέρημνας για τις ευαισθησίες στον γεωργικό μας τομέα. Και δεν θα πρέπει να έχουμε αυταπάτες γιατί η συμβολή τη Ευρωπαϊκή Γεωργία στι διαπραγματεύσει θα είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία ώστε το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων και από πολιτική και από οικονομική άποψη να γίνει αποδεκτό στους Ευρωπαίους Γεωργούς. Και το μήνυμά μου σήμερα είναι να κρατήσετε στενές επαφές με τους συναδέλφους στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και τους ενδιαφερομένους και τους ψηφοφόρους σας, ώστε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας να αντικατοπτρίζονται δεόντως στις γενικές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις διαπραγματεύσεις για το TTIP. Να πω λίγα λόγια και για τις γεωγραφικές ενδείξεις, που είναι προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις μας για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Βλέπετε με ποιες χώρες έχουμε συμφωνίες για γεωγραφικές ενδείξεις, είτε ευρεία είτε περιορισμένη και που διαπραγματευόμαστε το θέμα αυτό στο μέλλον. Οι γεωγραφικές ενδείξεις, όπως ακούσαμε, είναι ε, εμβληματικές μας εξαγωγές, είναι ε, εξαγωγές εμβληματικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ένταση απασχόλησης, απασχολούνται χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικροί καλλιεργητές και παραγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι γεωγραφικές ενδείξεις δεν είναι πια ή δεν είναι μόνο το προνόμιο λίγων κρατών μελών γιατί όλα τα κράτη-μέλη πια ε, προστατεύουν τα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη. Και όπως είπε ο κύριος Βίλσακ, η δεν ειναι μονο το προνομιο λιγων κρατων μελων γιατι ολα τα κρατη μελη πια προστατευουν τα προιοντα με γεωγραφικη ενδειξη και οπως ειπε ο κ. βιλσακ η φημη μας στην Ευρώπη ε, μιλάει για ποιοτικά, θρεπτικά, υγιεινά προϊόντα και από αυτήν την άποψη πρωτοστατούν εδώ τα προϊόντα γεωγραφική ένδειξη. Και γι' αυτό θα ε, εξασφαλίσουμε υψηλή προστασία στο TTIP για τι γεωγραφικές μα ενδείξει. Και σίγουρα η πρόταση που ακούσαμε από τι ΗΠΑ ε, δεν αρκεί. Δεν εξασφαλίζει την τέζουσα προστασία για τα προϊόντα μα που καλύπτονται από γεωγραφικέ ενδείξει. Θέλουμε ενισχυμένη προστασία γιατί μέχρι τώρα η προστασία τους είναι απαγορευτική, κυρίως για τους μικρούς γεωργούς και παραγωγούς μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, γιατί δεν αρκεί η διαπραγμάτευση για τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, θα πρέπει να ωφελούν αυτές με την πλήρη τους εφαρμογή τους γεωργούς μας. Γιατί υπάρχουν πολλοί φραγμοί, κυρίως υγειονομικών και φυτοϊγειονομικών προτύπων με τις τρίτες χώρες. Και αν υπάρχουν μη δοσμολογικοί φραγμοί τύπου υγειονομικών και φυτογειονομικών προτύπων, πάλι εμποδίζονται οι εξαγωγές μας. Οπότε και το θέμα αυτό μας ενδιαφέρει και μετά το ρωσικό εμπάργο, αλλά και ούτως ή άλλως θέλουμε να διαφοροποιήσουμε τις αγορές μας, αγορές εξαγωγής και να δούμε τι άλλα τι άλλα μη δημογραφικοί φραγμοί υπάρχουν, τύπου SPS. Ε, μετά από 15 χρόνια επαναφέραμε το κρέας μας στον Καναδά, γιατί εξαιτία τη πογκόδους κεφαλοπάθης είχαμε πρόβλημα, το ίδιο και με την Τουρκία. Και πολύ γρήγορα θα φτάσουν τα αχλάδια και τα μήλα μας και στην ε, Αμερικανική αγορά, να μένουν ε, η δημοσίευση των σχετικών διατάξεων. Και το ίδιο ισχύει για τη Λατινική Αμερική, γιατί εκεί υπάρχουν πολλές πολύ μη δεσμολογική φραγμή. Άλλη διάσταση του θέματο αφορά την πολιτική τη διαφημής τη πρόθεση μα και οι εμπορικέ μα αποστολέ στι διάφορε χώρε του κόσμου. Πρόσφατα με τη βοήθειά σας ε, εγκρίθηκε ο νέο κανονισμό για τη διαφήμιση, για την πρόωθηση μάλλον των προϊόντων που θα μπει σε ισχύ νουπο και όλο και περισσότερα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τον προπολογισμό και τι σχετικέ δραστηριότητε τη προώθηση των προϊόντων και διευρύνοντας ε, το καλά των προϊόντων στις ε, εκστρατείες ενημέρωση στον κόσμο. Και δεν στοχεύουμε στους ε, συνήθεις μόνο εταίρους μας, στους πιο γνωστούς, Κίνα, ΙΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες Αφρικής, Λατινικής Αμερικής και ούτω καθεξής. Και έχουμε και πολλές αντιπροσωπείες, αποστολές υψηλού επίπεδου σε διάφορες χώρες του κόσμου με συμμετοχή προσώπων των γεωργών, των παραγωγών από διάφορους τομείς. Τέτοιες αποστολές θα πραγματοποιηθούν το Φεβρουάριο στην Κολομβία και το Μεξικό, η Ιαπωνία, Κίνα τον Απρίλιο και Βιετνάμ και η Ινδονησία αργότερα το χρόνο και κατά πάσα πιθανότητα και στη Δυτική Αφρική. Πρόκειται για πολύ σημαντικές αγορές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Και βλέπω από τις αντιδράσεις ότι πρέπει να βάλω τελεία κάπου. Τώρα, για θέματα επιστημιστικής ασφάλειας. Πολύ εύγλωτα ο Υπουργός Βίλσακ μας μίλησε ότι μέχρι το 2050 θα πρέπει να θρέψουμε 9 δισεκατομμύρια κόσμο. Και μάλιστα ε, επειδή ακριβώ ε, η κατανάλωση θερμιδική αυξάνεται, είναι σαν να πρέπει να θρέψουμε 11 δισεκατομμύρια το 2050 και όχι απλώ 9. Μεγάλες επιστημιστικές ανάγκες θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε αλλά πιστεύω ότι με τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα το γεωρικό μα μοντέλο και να μοιραστούμε τι εμπειρίε μα και με του άλλου εταίρου μα, προκειμένου να έχουμε ισορροπημένη ανάπτυξη πέθρου, να βελτιώσουμε τον ε, εμπορικό προσανατολισμό των προϊόντων ώστε να αποφύγουμε στρεβλώσει ανταγωνισμού, να αναβαθμίσουμε τη κλίμακα αξιών με πιο ποιοτικά προϊόντα, να ε, επικεντρωθούμε και σε θέματα έρευνας και καινοτομίας και να προωθήσουμε την ανανέωση των γενεών στη Γεωργία. Και ο ρυθμός με τον οποίο θα εφαρμόσουμε αυτά τα θέματα θα επηρεάσουν όχι μόνο το επιστηστικό μέλλον της, Ευρω... Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Γιατί και η Ευρώπη αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις με τις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου. Επίτροπος στο επιτελείο του και η Γενική μας Διεύθυνση δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε σωστές επιστηστικές πολιτικές, από κοινού με τους εταίρους μας και αυτό το επιδιώκουμε στο G20, στο G7, στη ΦΑΟ, στη σχέση μας με την υποσαχάρια Αφρική και στην εφαρμογή των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας μετά το 2020. Οπότε η πολιτική μας δεν αφορά μόνο το εμπόριο και τις επενδύσεις, αλλά και την διάδοση καλών πολιτικών επιστηστικής ασφάλειας και πέραν των συνόρων μας. Και τέλος ήθελα να πω ότι προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Γεωργίας για να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες, να διευρύνουμε το εμπόριο, να ανοίξουμε τις αγορές και να αναπτύξουμε την εμπορική μας πολιτική με ισορροπημένο τρόπο σε συνεργασία με τους γεωργούς και με τους υπόλοιπους ενδιαφερμένους αλυσίδας ε, εφοδιασμού αξιοποιώντας τις ε, εμπορικές ευκαιρίες, αλλά προστατεύοντας ε, και τα αμυντικά μας συμφέροντα. Περιμένω λοιπόν και τη δική σας βοήθεια, ώστε οι ε, γεωρικές ευαισθησίες που έχουμε σε πολλούς τομείς να γίνουν αντιληπτές και στους εταίρους μας και να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές μας και τις στρατηγικές μας, είτε εθνικές είτε ευρωπαϊκές και στις διαπραγματεύσεις που έχουμε διεθνώς. Λυπούμε λοιπόν, που μακρηγόρησα, αλλά πραγματικά το θέμα είναι τεράστιο. Σας ευχαριστώ. Σας υποσχόμαστε πάντως ότι θα επαναρχόμαστε όλο και πιο συχνά στο θέμα αυτό. Δεν πρόκειται να εξαντλήσουμε σήμερα τη συζήτηση. Θα επαναρχόμαστε συστηματικά στο θέμα αυτό για να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγες την εξέλιξη των εμπορικών μα διαπραγματεύσεων και συμφωνιών. Και Σα υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε σχετικά σύντομα σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και έχουμε και μια παράκληση να έχετε πολύ σύντομε, μονόλεπτε παρεμβάσει γιατί πραγματικά δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Πρώτο ο κύριο Νίκολσον. Ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Νίκολσον. Uh, Καταρχά να σα διαβεβαιώσω ότι σίγουρα καλά τα καταφέρατε παρόλο που ακολουθήσατε το δύσκολο έργο του Αμερικανού Υπουργού Γεωργίας. Γίνουν διαπραγματεύσεις λοιπόν στον ΠΟΕ. Ερώτηση. Ο ΠΟΕ δεν πέθανε. Μόλις τις άλλες διαπραγματεύσεις που γίνονται, τι, τι, παναφερθήκατε στην Αυστραλία, το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία. Και είμαστε και νέοι ίσως ε, και άπειροι στις διαπραγματεύσεις αυτές που γίνονται στην Ευρώπη. Θα είναι σχετικό θέμα ο ΠΟΕ με τις διμερείς ε, συνομιλίες. Επέστρεψε στην ατζέντα στο Μέρκοσούρ μετά την πρόσφατη αλλαγή κυβέρνηση. Πρέπει να ανησυχούμε γι' αυτό. Με ισοδυναμίες. Πού βρισκόμαστε. Μυρίσαμε για εμπορικά σήματα και είπα υπερασπίστηκαν τα εμπορικά σήματα και το ανάφεραν. Θετικές ισορροπίες εμπορικές. Εντυπωσιακά αυτά. Αλλά αυτή η ισορροπία έχει τίμημα. Με τις διακυμάνσεις των τιμών όσον αφορά τις παγκόσμιες αγορές, πώς μπορούμε να κινηθούμε για να πετύχουμε σωστή ισορροπία. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά που προσήλθατε σήμερα ενώπιον μας σύντομη ερώτηση. Πού και πότε θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων για την TTIP. Και χαίρομαι επίσης που οι γεωγραφικές ενδείξεις εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα. Δεν είναι δυνατόν, αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον, δεν είναι δυνατόν να εγκαταληφθούν η συμφωνία περιλαμβάνει και ένα δεύτερο μέρος στο οποίο δεσμεύονται οι ΗΠΑ να δεχτούν και άλλες γεωγραφικές ενδείξεις εκτός από αυτές που είχαν εγκριθεί το 2006. Ο κ. Ντόρφμαν, γεωγραφικές ενδείξεις και εγώ. Είπατε, κ. Γενική Διευθυντά, ότι εδώ ανοίγονται ευκαιρίες για μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Όταν εξετάζω ποιος εξάγει αλλού στον κόσμο ε, ε, προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις βλέπω πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που εξάγουν. Δεν απαντήσατε καθαρά. Το ερώτημα δεν είναι αν έχουμε ίσα ή ισότιμα συστήματα. Το ζήτημα είναι εάν οι Αμερικανοί θα δεχτούν να χρησιμοποιήσουν τους δικούς μας χαρακτηρισμούς. Αν θα το κάνουμε αυτό με trademark ή με κάπως αλλιώς δεν είναι αυτό το θέμα δεν επιτρέπεται να επιτρέψουμε με τη σειρά μας να χρησιμοποιηθούν οι δικές μας γεωγραφικές ενδείξεις και από άλλα μέρη του κόσμου. Εδώ πρέπει να εξευρεθούν κάποιες λογικές λύσεις. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να επιτρέψουμε η TTIP να κατέλθει κάτω από το επίπεδο της συμφωνίας με τον Καναδά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριο Νταντάν. Ευχαριστώ. Δεν θα διέφυγε από πολλούς πριν ότι ο Υπουργό Γεωργία δεν απάντησε στην ερώτησή μου για τον ΠΟΕ και βλέποντας τον χάρτη των συμφωνιών στους οποίους συμμετέχουμε και πώς εξελίσσεται ο προπολογισμό της Βραζιλίας για τη Γεωργία της Ινδίας κλπ. και πως ποιες δράσεις διατίθεται, δεν πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα πλέον είναι όλο και πιο μόνη σαν θεματοφύλακας και προστάτης του ε, ναού που μιλώντας για αυτό το, το ναό αναφέρομαι στο ΜΠΟΕ και στην συμφωνία του Μαρακές. Κύριος Χάσλικ. Ο κύριος κάθε φορά σας βλέπουμε μας λέτε ότι τα πράγματα πάνε καλά και θα πάνε καλύτερα. Γιατί όμως τότε όσο ε, μεγαλώνει, διευρύνεται η παγκόσμια αγορά, μειώνονται οι τιμές των παραγωγών βλέπετε και τι γίνεται και με το γάλα. Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά. Και κάθε φορά που έρχεστε ξαναρχίζετε από την αρχή. Πεστε μου καλύτερα με ποιες χώρες δεν θέλετε να συνάψετε συμφωνία. Διαρωτώ με αν έχετε μια συνολική επισκόπηση γιατί με όλες αυτές τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που ε, διαπραγματεύεστε πώς θα εξασφαλίσετε τα ε, συμφέροντα των Ευρωπαίων Γεωργών Βεβαίω οι συμφωνίε περιλαμβάνουν και άλλα κεφάλαια και τα γεωργικά προϊόντα είναι αυτά, η γεωργική οικονομία είναι αυτή που επωφελείται λιγότερο από τι συμφωνίε. Και εν τέλει πρόκειται για ξεδιατροφιά. Κάθε φορά λέτε ότι θα διεξαχθεί συζήτηση. Και μα λέτε να έρθετε σε επαφή με του συναδέλφου σα τη Επιτροπή. Ίντα. Όχι, εγώ θέλω να συζητηθεί εδώ. Δεν θέλω απλώς να με εμφανίζετε το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών που έχουν γίνει αλλού. Ο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, ακούγοντάς σας, ενδυσηματίστε ότι τα πάντα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει πρόβλημα και εκπλήσωμα. Έχω μια ερώτηση αφορά τι ζωγραφικέ ενδείξεις. Ποια συγκεκριμένη είναι η πρόοδος της διαπραγματεύσεις όσον αφορά τι ζωγραφικέ ενδείξεις με τη ΣΥΠΑ. Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μας είπε ο υπουργό. δεν είναι προφανές ότι προχωρούν. Και αμφισβητείται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις γραφικές ενδείξεις. Η Γενική Διεύθυνση όσον αφορά, η αρμόδια, και για τα μη γεωργικά προϊόντα τις γραφικές ενδείξεις αν υπάρχει ε, κάποια πρόοδος. Η κυρία Σένερα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Έχω πολλές ερωτήσεις. Πρώτα. Με ποια ευρωπαϊκή ε, οργάνωση γεωργών θα πραγματοποιηθεί τις αποστολές, γιατί είπατε συμμετέχουν και πρόσωποι για γεωργών. Ποιας οργάνωσης. Μιλήσατε για τη συμφωνία με τον Καναδά. Εγώ ξέρω ότι δεν έχει τεθεί ακόμη σε σχέση. Όπω μα τα είπατε, σαν έχει ήδη εφαρμοστεί. Επίσης, ποια είναι τα ευαίσθητα προϊόντα ή ποια προϊόντα θεωρείται ευαίσθητα στις διαπραγματεύσεις του TTIP και για τα οποία δεν θα ανοίξουν πλήρως οι εισαγωγές. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπόγκοβιτς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Επιτροπή μας εγκρίναμε ένα ψήφισμα και μία έκθεση για το TTIP όπου λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι γεωργικές πρακτικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα. Έχω την αίσθηση ότι δεν γίνονται σεβαστές οι χείουσες πρακτικές αλλά προσπαθούμε να μπούμε στο καλούπι των αμερικανικών πρακτικών στο θέμα των φυτοφαρμάκων. Κάτι που αφήνει ανυπεράσπιστους ε, τους Ευρωπαίους γεωργούς και τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Είναι πολύ ευάλωτη η γεωργοί μας απέναντι σε αυτήν την κατάσταση και θα έπρεπε κανονικά να τύχουν περισσότερης προστασίας. Γιατί με τα μέτρα αυτά θα γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν την προστασία της ε, γεωργικής καλλιέργειας και παραγωγής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φαίνεται παράξενο αλλά τελικά θα λείπουν πολλά προϊόντα, θα έχουμε λήψει σε πολλά προϊόντα, αυξάνεται ο πληθυσμό, μακροπρόθεσμα θα γίνει αυτό, αλλά εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε πλεόνασμα γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατο. Επενδύαμε στι νέε αγορέ και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τι, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν είναι αρκετά καλές οι αγορές. Γιατί δημιουργείται το πρόβλημα. Ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος της συμφωνίας με τις Πολιτείες. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πολλές μελέτες λένε ότι η αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα επηρεαστεί αρνητικά από τη συμφωνία και ότι θα έχουμε αρνητικό πρόσημο όσον αφορά την ισορροπία. Θα είναι αρνητικό το αποτέλεσμα. Η δική σας αντίδραση ποια είναι. Κυρία Γιλέρα, ευχαριστώ. Έχω δύο πολύ Συγκεκριμένε ερωτήσει προ τον, πρόεδρο της στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκατε στη συμφωνία με το Βιετνάμ που έχει προβληματίσει τα μάλα τους ριζοκαλλιεργητές της Ανταλουσίας και της Ισπανίας γενικά. Τι γίνεται, ποια είναι η θέση των Ευρωπαίων ριζοπαραγωγών για τη συμφωνία με το Βιετνάμ. Μπορείτε να το διευκρινίσετε. Και ξεχάσετε λίγο στα προκυβευτικά, το ελαιόλαδο, που είναι πολύ σημαντικά προϊόντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη. Με τις συμφωνίες αυτές ε, θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για τα προϊόντα αυτά ή μήπως ε, θα ζημιωθεί η παραγωγή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιθυμώ να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς ορίζει τους ευαίσθητους τομείς. Θα ήθελα να ακούσω από εσάς θίξατε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τις εμπορικές συμφωνίες. Αφενός το γάλα, όπου οι ΗΠΑ αύξησαν τους δασμούς για προϊόντα βουτύρου και ε, κρέμας, σαν τη γη κτλ. Από την άλλη μεριά, τα αμύγδαλα της Καλιφόρνιας που παράγονται με χρήση μεγάλοι ε, ζανιοκτών και έχουν ε, εξαφανιστεί οι μέλισσες από την περιοχή αυτή, πώς θα προστατεύσετε εσείς την ευρωπαϊκή καλλιέργεια αμυγδάλων. Μιλάτε και για πολλά πλεονεκτήματα δήθεν υπέρ της ε, αγροτικής οικονομίας. Εγώ βλέπω περισσότερα πλεονεκτήματα να αποκομίζει τελικά η μεταποιητική βιομηχανία τροφίμων, όχι όμως οι γεωργοί και οι αγρότησες. Κύριε Κλάρκ εντάχει μια ερώτηση. Στη συμφωνία του Ειρηνικού, είπα, με 11 χώρες πέτυχαν λοιπόν όσον αφορά συγκεκριμένη σημασία για τις γραφικές ενδείξεις. Είναι επικίνδυνη αυτή η συμφωνία ή όχι όσον αφορά εμάς. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ. Σε σχέση με τα σχόλιά σας και σχόλια άλλων για τα όσα είπε ο Υπουργό Γεωργία στον ΗΠΑ. Όταν θε να κάνει μια συμφωνία με κάποιον, πρέπει να είσαι φιλικό όταν θε να συμφωνήσει. Λοιπόν, νόμιζα ότι πολλοί πολλά από αυτά που μα είπε ήταν ενδιαφέροντα, αλλά δεν μα ενέπνεαν. Και αναφέρθηκε στο όταν ήταν κυβερνήτη. Όταν ήταν κυβερνήτη θεωρήθηκε από την ε, ε κυβερνήτη τη χρονιά για βιοτεχνολογικά προϊόντα. Και αυτό θα με ενοχλούσε. Δεν είναι και τόσο ή ε, ήπιος ε, και γλυκός όπως θεωρούμε. Διότι αν πήρε εκείνο το βραβείο τότε το πήρε για κάποιο λόγο. Ο νόμος που ανέφερα ξεκίνησε το νομοσχέδιο. Ήθελε να πάει να τον ξαναδιαβάσει το νόμο και αυτό με ανησυχεί διότι διαπραγματευόμαστε μαζί τους και οι διαπραγματεύσεις και που βλέπω είναι συνέχεια να τον κολακεύουμε. Και ποιος διαπραγματεύεται από την άλλη πλευρά. Ο Φιλ Χόγκαν κάποιος που περιγράφεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Γαλακτοπαραγωγών ότι δεν έχει λύσεις, ότι δεν είναι ικανός επαγγελματικά και αγνοεί τους γεωργούς. Εγώ τρέμω στην ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά θα πάει να διαπραγματευτεί με κάποιον εδώ που είχε περιγραφεί σχεδόν σαν να ήταν ο Ιησούς όταν έφυγε από εδώ. Δηλαδή τον, πολύ τον λατρέψαμε τον Υπουργό. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Γενικό Διευθυντή. Εγώ είμαι υπέρ της εταιρικής σχέσης. Ταξιδεύω συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες και βλέπω και με τα μάτια μου τις ευκαιρίες που θα έχουν οι Ευρωπαίοι Γεωργοί από τις συζητήσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πέραν των γεωγραφικών ενδείξεων μιλήσατε καθόλου για την σήμαση των προϊόντων. Γιατί ξέρω ότι στην Ευρώπη έχουμε προβλήματα με την σήμανση των προϊόντων σε σχέση με τη χώρα προέλευσης. Μάλιστα είχαμε εγκρίνει και σχετικό ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι διχασμένο. Για τις χώρες προέλευσης μπορούμε να μιλήσουμε στις διαπραγματεύσεις ε, κυρίως για τα προϊόντα που έχουν ως βάση το κρέας. Ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε η Ρωσία αποφάσισε να απαγορεύσει εισαγωγές από τις δυτικές οικονομίες. Οι καταναλωτές τους όμως θα εξακολουθούν να θέλουν φαγητό. Διερωτώ με, οι έρευνες που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δει δείξει ότι έχουν αυξήσει οι εξαγωγές προς Λευκορωσία, Ουκρανία, Καζακστάν από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσης και άλλες πρώην Σοβιετικές χώρες που είναι μουσουλμανικές και προς την Μογγολία. Άρα υπήρχε κάποια εξαγωγή από την πίσω πόρτα που έγινε προς τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, παρακαλώ, σύντομα να απαντήσετε και αν ε, δεν προλαβαίνετε ή δεν ε, είστε έτοιμος μπορείτε να στείλετε και γραπτός απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Σημείωσα ότι κάλυψαν περίπου 7 θέματα. Ο ΠΟΕ πέθανε, βέβαια δεν πέθανε. Ο ΠΟΕ όχι μόνο είναι διαπραγματευτικός φορέας, αλλά και φορέας ο οποίος παρακολουθεί την εφαρμογή των εμπορικών κανόνων. Είναι καθημερινή του δουλειά και απειλή και διαφορές εμπορικής φύσης. Ακόμα και αν τα θέματα, οι διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά στον ΠΟΕ έχουν αποτελματωθεί, για να το πω έτσι, σε αυτή τη φάση, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να είναι αντικείμενα διαπραγματεύσεις μόνο στον ΠΟΕ. Παραδείγματο χάρη, κανόνε για κάποιε επιδοτήσει όπω την Αλία ε, δεν μπορεί να τα διαπραγματευτεί κανεί δίμερος Πάντα λοιπόν θα υπάρχει περιθώριο στα πλαίσια του ΠΟΕ για τη διαμόρφωση κανόνων εμπορικών. Ακόμα και αν το θεματολόγιο υπόσχεση στην αγορά έχει ξεπεραστεί κάπως από την διάδοση ελεύθερη των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου που συνάπτονται στον κόσμο. Κάτι αναφέρθηκε επίσης για το επίπεδο της στήριξης που στευλώνει την αγορά από τις αναδυόμενες οικονομίες γίνεται αυτό. Πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση από εκεί που ε, ε, στήριζε το πράσινο τετραγωνίδιο η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία κινούνται προς την αντίθετη ε, κατεύθυνση. Στηρίζουν τους γεωργούς και αυτό πρέπει να διευθετηθεί στη διαπραγματεύση των ΜΟΕ κατά πόσο στρεβλώνεται η αγορά είτε όχι. Άλλες ερωτήσεις για το TTIP, επόμενος γύρος δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Ίσως ε, τέλος Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου ε, στις Βρυξέλλες η αρχες φεβρουαριου στις βρυξελλες η δεν, η σήμανση δεν συζητήθηκε σε αυτή τη φάση του TTIP. Οι ΕΠΑ θέλουν να εκμεταλλευτούν ή να διαρευνήσουν την χρήση της σήμανσης για να δώσουν επιλογή στους καταναλωτές. Πράγματος χάρη γενετικά τοπημένα προϊόντα, μη γενετικά τοπημένα προϊόντα δεν είναι κάτι που υποστηρίζουμε στην Ευρώπη διότι έχουμε απλώς απαγόρευση όσον αφορά τις ορμόνες και την παρουσία γενετικά τουμένων οργανισμών, άρα η σήμανση δεν λύνει το πρόβλημα για μα. Ε, ερώτηση. Ποια είναι τα ευαίσθητα προϊόντα στι πραγματεύσει TTIP και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Αναφέρθηκα σε κάποια από αυτά. Δεν διατείνομαι ότι κάλυψα όλες τις ευαισθησίε, αλλά είναι σαφέστατο ότι το βόιο, τα πουλερικά, το χείριο και ίσως όχι το πολύ κατεργασμένο χείριο, αλλά βασικά προϊόντα χειρίου ε, εθανόλη, ζάχαρη, άμυλο. Ε, όλα αυτά είναι αρκετά ευαίσθητα προϊόντα αντί τον είπα. Στι περισσότερε περιπτώσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οικονομία κλίμακα δεν είναι τόσο καλή. Η μείωση, ε, το κόστος παραγωγής είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι της είπα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε υψηλή δασμολογική προστασία. Και οι ποσοστώσει τα προϊόντα, για τα ευαίσθητα προϊόντα δεν θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε πλήρως τις αγορές. Κάποιοι αναφέρθηκατε σε πρόσφατη μελέτη που έγινε από την Υπουργείο Γεωργίας τον ΗΠΑ που υπολόγισε ότι αν απελευθερώναμε πλήρως όλα τα προϊόντα μας οι ΗΠΑ θα κέρδιζαν 5,8 δις δολάρια όσον αφορά τη βελτίωση εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς θα κερδίζαμε μόνο 0,8 εκατομμύρια σε περισσότερες εξαγωγές προς τη ΗΠΑ και με πλήρη απελευθέρωση του βοήου θα είχαμε 1,1% μείωση στον όγκο της παραγωγής και των τιμών στην Ευρώπη. Πλήρης απελευθέρωση λοιπόν δεν θα ήταν εφικτή, θα πρέπει να δούμε για ποσοστώσεις δασμολογικής μείωσης για να δώσουμε καλύτερη πρόσβαση στη ΣΥΠΑ και να βρούμε λύση. Τώρα, οι ονομασίες προέλευσης, οι γεωγραφικές ενδείξεις που θίξατε πολύ, εγώ δεν συμφωνώ ότι είναι κάτι που αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις ακόμα και τα περισσότερα σημαντικά ονόματα όπως είναι το Παρμεντζάνο Ρετζάνο με ονομασία προέλευσης αυτό το όνομα, αυτό, αυτή η εταιρεία απασχολεί, αυτό το όνομα απασχολεί 50.000 ανθρώπους σε εκμεταλλεύσεις, συνεταιρισμούς κλπ. σε αυτό το τμήμα της Ιταλίας. Οι περισσότερες ονομασίες προέλευσης μπορούν να δούμε ότι ανήκουν σε πολύ μικρές παραγωγές και σε πραγματεύσεις με τον ΙΠΑ προτείναμε να προστατεύσουμε καλύτερα περίπου 250 ονομασίες συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι αρκετά μέτρες επιχειρήσεις όπως προυνόνταυσαν ε, ε, ή συγκεκριμένο αχλάδι ε, από την Πορτογαλία, του Ρόντα, Λικάντε κλπ. Διάφορα τέτοια προϊόντα πίσω κρύβονται μικροί συνεταιρισμοί, μικρή παραγωγή πίσω από αυτά τα ονόματα των προϊόντων. Κάποιο ρώτησε τι γίνεται συμφωνία για τον Ίνο του 2006. Σε αυτή τη συμφωνία είχαμε προστατεύσει αρκετά, αρκετούς ίνους και είναι και από τις δύο πλευρές, αλλά είχαμε αφήσει κάτι εκρεμές για τα ινή γενώσιμα, πόρτο και σαμπάνια και διάφορα άλλα και είχαμε ε, ρήτρα αναθεώρησης που θα, εκεί που θα διαπραγματευόμαστε την οριστική λύση για τα ονόματα ή τις ονομασίες αυτές. Οι ΙΠΑ δεν ήταν ποτέ έτοιμες να αντιμετωπίσουν τη σταδιακή εξάλληψη του μέτρου αυτού των ημιγενοσύμων, οπότε μόνο μέσω των TTIPs, του TTIPs μπορούμε να λύσουμε αυτό το θέμα και να προστατεύσουμε τα, τα 17 πολύ σημαντικά ονόματα ενοπνευματοδών και ίνων της Ευρώπης, ισοδυναμία συστημάτων. Ε, δεν νομίζω ότι το σύστημα εμπορικών σημάτων των ΗΠΑ παρέχει επαρκή λύση για να προστατεύουμε τις, ε, τις ευρωπαϊκές ονομασίες προέλευσης για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν παρέχεται το υψηλό επίπεδο προστασίας που απαιτείται για τα τρόφιμα και δεύτερον το κόστος επιβολής της ονομασίας στην αγορά της, ε, των ΗΠΑ ε, με εμπορικό σήμα είναι απαγορευτικό σε ύψος για τις μικρές εταιρείες. Εκατομμύρια δολάρια κοστίζει ε, συνεχώς προσπάθειες για να επιβάλλεις την ονομασία σου στην αγορά. Αυτό που επιδιώκουμε είναι, χωρίς να ζητάμε από τις ΣΥΠΑ να θετήσουν το δικό μας σύστημα ονομασιών προέλευσεως, να βρούμε έναν άλλο τρόπο να πετύχουμε προστασία των ονομασιών των προϊόντων στην αγορά των ΗΠΑ. Στις συμφωνίες της ΗΠΑ δίνει προστασία σε ονομασίες προέλευσης στα ενοπνευματόδη, όπως το whisky, του Tennessee και το bourbon. Ε, τα θεωρεί διακεκριμένα προϊόντα και σε συμφωνίες παρέχει προστασία για αυτά τα διακεκριμένα προϊόντα. Ε, είναι κάτι άλλο πέρα από ονομασία. Είναι ε, σχεδόν προστασία ονομασίας προέλευσης. Μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς να χρησιμοποιήσουμε την προστασία ε, μέσω εμπορικού σήματος των ΙΠΑ, ε, να χρησιμοποιήσουμε ένα ιδιαίτερο σύστημα. Δεν έχουμε πετύχει πρόοδο στον αφορά τις ονομασίες προέλευσης με τις ΙΠΑ, είναι πολύ δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, όμως αναγνωρίζουν οι ΙΠΑ ότι θα πρέπει να υπάρξει στο τίτυπο αποτέλεσμα για τις ονομασίες προέλευσης, η γεωγραφική ονομασία, αλλιώς δεν θα περάσει η συμφωνία από το Συμβούλιο, από το Κοινοβούλιο και να γνωρίζει την ΙΠΑ ότι δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε σε αυτού ή να επιβάλλει ο ένα τον άλλον το σύστημά του. Αυτό είναι μια πρόοδος, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μα. Ένα, κάνας δύο είπατε ότι θεωρούσα ότι ήμουν πολύ αισιόδοξο και αφελή όσον αφορά τι μελλοντικέ διαπραγματεύσει. Προσπάθησα να πω ότι έχουμε πραγματικά προβλήματα μπροστά μας όσον αφορά το δομέα του κρέατος και άλλους τομείς, δοθέτως ότι τώρα είμαστε θα συναγωνιστούμε με τον Καναδά, με πιο ανταγωνιστικές οικονομίες. Έχουμε τη ΣΥΠΑ, Μερκοσούρ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Πολύ ανταγωνιστική. Πρώτα απ' όλα δεν θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε πλήρως ε, τους βασικούς τομείς και δεύτερον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το σύνολο των διαπραγματεύσεων σφαιρικά τόσο ώστε να μην θετήσουμε κατακαιρματισμένη προσέγγιση τμηματική και να προσφέρουμε χωρίσεις ε, έτσι ε, σε διάφορους τομείς και διάφορες επαγματεύσεις να λαμβάνουμε υπόψη τη ε, συνολική εικόνα. Μερκοσούρ ίσως ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο Εμπορίου το συζητήσαν και δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε ποιο επίπεδο θα συνεχιστούν. Λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις σε τα δεν ξέρουμε που βρισκόνται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα τεθεί αν εξαρτάται από τις αποφάσεις ποιο σύστημα ε, διευθετήσεως των διαφορών θα ενταχθεί στη συμφωνία αυτή. Βιετνάμ, ε, ανησυχίε για το ρύζι, ελαιόλαδο και φρούτα. Για το ρύζι προσφέραμε ε, κάποια ποσόστοση για το ρύζι, για απελευθέρωση της ποσοστώσης, σχετικά μικρό ποσοστό που δεν θα έχει αντίκτυπο όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά ή τις τιμές και για το ελαιόλαδο και για τα φρούτα και τα, και τα οποροκυπευτικά. Οι Βιετναμέζοι εξάγουν κάποια τροπικά φρούτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό με τη δική μα παραγωγή. Για το ελαιόλαδο έχουν απελευθερώσει πλήρω την ε, αγορά του. Λοιπόν, έχουμε εξαγωγικέ δυνατότητε για το ελαιόλαδο στο Βιετνάμ. Τελευταία δύο σημεία για τη συμφωνία του Ειρηνικού και για τη Ρωσία. Για τη Συμφωνία του Ειρηνικού υπάρχει ένα κεφάλαιο για τις γεωγραφικές προελεύσεις στη Συμφωνία, που δεν απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά αναφέρει όταν θες να προστατεύσεις νομασίες προέλευσης, γεωγραφικής προέλευσης, θα πρέπει να ακολουθήσεις μια διαδικασία σωστή, να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει δυνατότητα ε, ένστασης από ανταγωνιστικά συμφέροντα να πούν αν είναι εννοώσιμο, είναι μόνο εμπορικό σήμα, δεν είναι γεωγραφική ονομασία. Το κάνουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο κάνουν και εταίροι μα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, ε, δεν με εντυπωσιάζει το αποτέλεσμα αυτό που πέτυχαν εκεί στον αφορά τη Συμφωνία του Ειρηνικού για τη Ρωσική Ομοσπονδία τελικά ε, πράγματι, αυξήθηκε το εμπόριο από Λευκορωσία ε, προς τη Ρωσία και από τις Βαλκανικές χώρες, ίσως για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα ίσως να υπήρχε κάποια απάτη, ε, λάθος σήμανση, δεν ξέρουμε. Η Ρωσία συνεργάζεται με τις αρχές της Λευκορωσίας να δει κατά πόσο τίθεται αυτό το θέμα. Δεύτερον, δεν μπορέσαμε να εξάγουμε πλέον τυρί στην Ρωσία. Αυτό που συνέβη λοιπόν ήταν ότι η παραγωγή γαλακτοκομικών εξήγαγαν γάλα στη Λευκορωσία και η μεταποίηση σε τυρί έγινε στη Λευκορωσία και ίσως κάποιες άλλες χώρες και μετά νόμιμα εξήχθη ε, προς τη Ρωσία. Ε, είναι επιλογή επιχειρηματική αυτή να γίνει η μεταποίηση στη Λευκορωσία και τρίτον έγινε και κάποια αλλαγή μετακίνηση. Δεν εξάγουμε πλέον χείριο προς τη Ρωσία Οπότε άλλε χώρε τη περιοχή άρχισαν να καλύπτουν το κενό εξάγοντα χείριο στη ρωσική αγορά. Εμεί με τη σειρά μα εξάγαμε στην τρίτη χώρα χείριο η οποία εξήγαγε το προϊόν τη στη Ρωσία. Οπότε υπήρχαν διάφοροι τρόποι με του οποίου άλλαξαν οι μορφέ του εμπορίου και δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι κάποια σκοτεινή διαδικασία, κάποια σκοτεινή δραστηριότητα. Σα ευχαριστώ. Όπως ε, υποσχέθηκα θα επανέλθω στο θέμα αυτό σχετικά γρήγορα. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το 6. Παρακαλώ, ας έρθουν οι καλεσμένοι μας στην έδρα. Και εν τω μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι αμέσως μετά τις 6.30 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Γεωργών παραθέτει χριστουγεννιάτικη δεξίωση στο εστιατόριο που βρίσκεται στο κτίριο που βρισκόμαστε. Γιώζεφ Άνταλ. Ήθιστε κάθε χρόνο να μας προσκαλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Γεωργών σε χριστουγεννιάτικη δεξίωση που θα ξεκινήσει σήμερα στις 6.30 στο εστιατόριο που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο του κτίριου μας. Πάμε τώρα στην παρουσίαση της μελέτης ε, για τους συντελεστές της γεωργικής παραγωγής ή τις γεωργικές εισρωές. Το θέμα των ε, τιμών γεωργικών προϊόντων, την επιρροή τους ε, στα γεωργικά εισοδήματα, τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια στο κόστος της παραγωγής και τι γίνεται με την ενέργεια, τα, τους σπόρους, τα φυτοφάρμακα και πώς συμβάλλουν αυτά στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, ε, εμπειρογνώμονές μας, τον κύριο Γιώστος Βέσελερ και τον κύριο Ντούσαν Τράπικ από το Πανεπιστήμιο Βάγκενίγκεν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βέσελερ, που είναι ένας από τους ε, συντάκτες της μελέτης, για να μας κάνει την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με αισθάνομαι μεγάλη τιμή που θα σας παρουσιάσω τα πορίσματα της μελέτης μας. Τώρα ακουγέστε καλύτερα, λέει ο Πρόεδρος. Μπορείτε να επαναλάβετε. Βεβαίως, νιώθω μεγάλη τιμή που μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα τα πορίσματα της μελέτης μας για τη συγκέντρωση ε, και την επισκόπηση των γεωργικών ισορροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίμα που έμεινε για το τέλος ε, ε, της ε, συνεδρίασης. Μάλιστα στο Βάγκενινγκ στο Πανεπιστήμιο ε, σκεφτήκαμε να προτείνουμε να γίνονται μαθήματα και το απόγευμα προς το βράδυ, αλλά βλέποντα πόσο λίγοι έχετε μείνει στην αίθουσα, μάλλον θα καταπέσει τελικά αυτή η πρόταση για βραδινά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Βάγκενιγκεν. Να σας παρουσιάσω λοιπόν την έκθεση που στην μελέτη που υποβάλαμε με το επιτέλειο μου. Εγώ είμαι υπεύθυνο γεωργική και οικονομική πολιτική στο Πανεπιστήμιο Βάγκενινγκ και μαζί μου στο επιτελείο συμμετείχαν ο Αλεσάνδρο Μπονάνο και ο Ντούσαν Ντράπικ που κυρίω ασχολήθηκαν με τη ζήτηση και η Βαλεντίνα Ματέρια, Τόμα Βένου, Λούκα Μαλαγκούτη και Μάιερ με την υπόλοιπη μελέτη. Είχαμε εδώ τις αιτήσει αλλαγές κατά μέσο όρο των γεωργικών εισοδημάτων στην περίοδο 2004-2012 για μερικές χώρες και για διάφορους τομείς των γεωργικών εισρώων, για παράδειγμα σπόρους, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Βλέπετε ότι οι δαπάνες διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και οι τάσεις τους επίσης είναι διαφορετικές. Και αυτό μας δίνει κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τις συνέπειες και τον, τα επίπεδα συγκέντρωσης των γεωργικών συντελεστών. Βλέπουμε ότι είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση μεταξύ των κρατών μέλων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις σημαντικές διαφορετικές διαφορές που έχουμε στα κράτη-μέλη. Τώρα, γιατί χρειάστηκε αυτή η μελέτη. Γιατί είχαμε αύξηση στην αστάθεια σε ό,τι αφορά τις τιμές των πόρων. Γνωρίζουμε ότι οι συντελεστές αυτοί είναι σημαντικοί για τον γεωργικό κλάδο και είχαμε μια αύξηση του χάσματος μεταξύ των τιμών ισορών και ακρών στον γεωργικό τομέα. Για να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό χρησιμοποίησαμε δύο ε, βάσεις δεδομένων, το, ε, το FADN, το Standard Gross Margin Method και το Standard Output, Output Method. Και επίσης τα στοιχεία της Eurostat ε, τη Φάουστατ και συγκεντρώσαμε πληροφορίες και από ιστοσελίδες και επιστημονικά δημοσιεύματα. Είδαμε τη συγκέντρωση στη ζήτηση, τη συγκέντρωση στην προσφορά. Επίση αυτό που κάναμε είναι προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τι μορφή έχει η συγκέντρωση χρησιμοποιώντας τον δείκτη Herpindal-Hirschman. Αυτό είναι βασικό δείκτη συγκέντρωση. Θα ε, σε αυτό αργότερα. Για να δούμε του σπόρου πρώτα, το, το μέτρο σπόρων. Έχουμε το, κατα, τη μέση τιμή κόστου των σπόρων στα κράτη-μέλη. Βλέπουμε σημαντικέ διαφορέ ε, μεταξύ των κρατών μελών. Σε μερικέ χώρε οι δαπάνε για του σπόρου αυξήθηκαν, ενώ σε περισσότερε χώρε ε, οι δαπάνε αγορά σπόρων μειώθηκαν σταδιακά. Βλέπουμε εδώ τη συγκέντρωση στις 10 πρώτες εταιρείες ε, σπόρων. DuPont Pioneer, Monsanto και Syngenta είναι μεγαλύτερες, κατόπιν Limagren, KWS, Baker, Crop Science, Dow, DLF, Sakata και Land O Lakes. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες ε, εταιρείες. Και σε ό,τι αφορά τους συντελεστές συγκέντρωσης έχουμε μεταξύ 705 ε, και 673. Μικρή αύξηση μεταξύ 2000 10 και 12 και μετά μικρή μείωση. Τώρα γενικώ για την αγορά των σπόρων. Οι διαφορές είναι μεταξύ 2 και 15% μεταξύ των κρατών μελών. Είχαμε μια σταδιακή φθήνουσα πορεία. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι λιγότερο συγκεντρωμένη και η μέση συγκέντρωση είναι 673, σχετικά χαμηλή. Πάντως υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη συγκέντρωση μεταξύ των αγορών σπόρων. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την αγορά σπόρων ζαχαροτέφυλλου έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση της τάξης του 2444. Οπότε χρειάζεται κάποια προσοχή εκεί και σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις και τις αγορές βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά χαρακτηρίζεται περισσότερο από επενδύσεις και τεχνολογία παρά από αγορά εταιριών σπόρων. Και η αγορά εταιριών σπόρων από τις μεγαλύτερες 10 κυρίως συγκεντρώνεται στις ΗΠΑ. Σε ό,τι αφορά την αγορά ζωοτροφών βλέπουμε ότι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των γεωργικών εισρωών οι ζωοτροφές. Και εκεί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Σε ορισμένες χώρες οι αυξήσεις τις δαπάνες είναι μεγάλη, είναι σημαντικές, ενώ σε υπάρχουν μειώσεις. Πάντως θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση για τις ζωοτροφές μεταξύ των διαφόρων ειδών ζωοτροφών. Και επίσης ε, στο, στις συμπυκνωμένες ζωοτροφές και εκεί έχουμε στις 10 βασικότερες εταιρείε παραγωγή που ποικίλει μεταξύ 6,40 μεγατόνους ε, για τη μεγαλύτερη το 1 μεγατόνο για τις μικρότερες. Γενικώ 16% του συνολου... της συνολικής παραγωγής ζωοτροφών ε, παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει μεγάλη εμπορική κίνηση στον τομέα αυτό. Και η μεγαλύτερη παραγωγή είναι στη Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, κάτω χώρες, Βέλγιο και Πολωνία. Και ο τζίρος έχει αυξηθεί κατά 50% τα τελευταία 8 χρόνια, ενώ στις περισσότερες εταιρείες έχει μειωθεί κατά 15%. Άρα υπάρχει συγκέντρωση στον τομέα των ζωοτροφών. Όταν όμως βλέπουμε τους ε, λόγους της συγκέντρωσης, τους συντελεστές συγκέντρωσης, δεν μας ανησυχούν από οικονομική άποψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενέργεια, εκεί παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες στην ενέργεια έχουν αυξηθεί ε, στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Το μεγαλύτερο μερίδιο το φέρουν τα καύσιμα και ακολουθεί το φυσικό αέριο και κάποια άλλα ενεργειακά προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τους συντελεστές συγκέντρωσης, εκεί διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών κλάδων της ενέργειας. Αν το συγκρίνουμε με, άλλες, με άλλους γεωργικούς συντελεστές, βλέπουμε ότι η συγκέντρωση στην ενέργεια είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλους γεωργικούς συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν κατακλείδη, η γεωργία στην Ευρώπη έχει γίνει πιο ενεργειοβόρα και στις 23 από τις 27 χώρες μέλη πάνω από το 50% του κόστους ε, ενέργειας αφορά ε, ε, λιπαντικά και καύσιμα κινητήρα. Και έχουμε κυρίως κάθετη συγκέντρωση. Στην ενέργεια, επαναλαμβάνω, η συγκέντρωση αυξάνεται σταδιακά, κυρίως στο αργό πετρέλαιο. Έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση, κατόπιν φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα και από την υπόλοιπη τομή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα λοιπάσματα, και εκεί διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένε χώρε οι δαπάνε για τα λοιπάσματα έχουν αυξηθεί. Γίνεται όμως διαφοροποίηση μεταξύ των, του νητρογόνου φωσφάτου και ποτάσιου, πότας. Ε, κυρίως για νητρογόνα, ε, αζωτούχα έχουμε περισσότερες δαπάνες και βλέπουμε τις 10 μεγαλύτερες χώρες. Εκεί ε, μεσαία είναι η συγκέντρωση, 200 με 206 ο συντελεστής. Και η συγκέντρωση δεν έχει αλλάξει ε, εντυπωσιακά τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση έχει μειωθεί στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως διαφορές σε ό,τι αφορά τα ζωτούχα, τα καλλιούχα και τα φωσφατούχα. Και έχουμε μια σταδιακή αλλά ε, σχετικά φθήνουσα πορεία. Τώρα, τα τελευταία χρόνια είχαμε μείωση της, ε, των βελτιωτικών του εδάφους, ενώ η συνολική αξία των, των πωλήσεων ε, φυτοφαρμάκων έχει αυξηθεί στην περίοδο 2003-2012 και αυξήθηκε η πώληση βελτιωτικών εδάφους. Η Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ηνωμένα Βασίλειο και κάτω χώρε ε, αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού τζίρου λοιπασμάτων στι 27 χώρε. Μέτρια είναι η συγκέντρωση εδώ και μάλιστα ε, είχαμε αρκετέ συγχωνεύσει και αγορέ, αλλά μικρή η συγκέντρωση, μέτρια μάλλον. Τώρα σε ό,τι αφορά την, ε, τις, σε ό,τι δαπάνες για, για τη φυτοπροστασία έχει μειωθεί ε, ο συντελεστής. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τα διάφορα προϊόντα, πρώτα έχουμε ζενιοκτώνα, μετά Μεγιτοκτώνα και το καθεξής. Σε ό,τι αφορά τη, τους συντελεστές συγκέντρωσης, επικύλουν από 1556 ε, με 1717. Τώρα, η αξία των ε, της προστασίας των φυτών ε, έχει αυξηθεί μέχρι το 2008 και μετά άρχισε να πέφτει. Γενικώ υπήρχε μείωση στην όλη παραγωγή. Τα φυτο, φυτοκτόνα είχαν τα μεγαλύτερα ποσά, κατόπιν έχουμε τα μικητοκτόνα και στις μεσογειακές χώρες μεγαλύτερη ε, χρήση εντομοκτόνων και μικρότερη χρήση ζύζανιοκτόνων. Το συνολικό κόστος πάντως ε, το γεωρικό έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια για τις 15 παλιές χώρες, ενώ αύξηση έχουμε στις 10 νέες χώρες. Και σε ό,τι αφορά την προστασία των φυτών, είχαμε μείωση μέχρι το 2009 και αύξηση κατόπιν. Ο αριθμό των ε, εταιριών που παράγουν τέτοια φυτοπροστατευτικά προϊόντα μένει σταθερό. 630 με 655 είναι οι επιχειρήσεις και ο τζίρο είναι μεγαλύτερο στη Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Τώρα, ο κλάδος ε, προϊόντων φυτοπροστατευτικών έχουμε ένα σπάνικ από 79 μέχρι 83% Έχουμε μείωση του δίκτυ τα τελευταία χρόνια μετά από μία διακύμανση και αυτό εξηγείται από το υψηλό επενδυτικό κόστος της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Και τέλος, δεν έχουμε κάποιο ξεκάθαρο πρότυπο σε ό,τι αφορά την ζήτηση σημαντικών τέτοιων τομέων γεωργικών εισρώων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη συγκέντρωση η ορατή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τις γεωργικές εισρωές. Με εξαίρεση τα, τις οτροφές όπου έχουμε 65% στη, ε, στη Μάλτα, ε, αλλά στις περισσότερες χώρες κάτω από 35%. Κάτω από 30% μάλλον. 13% στη Λιθουανία. Έχουμε μεγάλες διακοιμάσεις. Πάντως, ε, αν λάβουμε υπόψη τη συγκέντρωση, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ζωτροφές. και έχουμε τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Και αυτή είναι μια σύνοψη της ζήτησης βλέπουμε τις τάσεις για τους σπόρους. Φθήνουσα απορία, αύξα, απορία πορεία στους ζωοτροφές, ε, σχετική μείωση στην ενέργεια και στα φυτοφάρμακα και τη φυτοπροστασία σχετικά σταθερά επίπεδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές συγκέντρωσης για την προσφορά, έχουμε τη μεγαλύτερη ε, προσφορά στο θέμα της φυτοπροστασίας από τις γεωργικές ροές και τη λιγότερη συγκέντρωση ε, στα φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, συγγνώμη, και τις ζωοτροφές. Αυτά εγώ τελείωσα και περιμένω τις απορίες σας. Ποιο θέλει το λόγο, παρακαλώ. κύριος Άγνιου ζήτησε το λόγο. Θέλω να μου πείτε ποιος άλλος θα ενδιαφέρεται για να μπορέσω να σας μοιράσω το χρόνο αγόρευσης. Ο κύριος Άγνιου, κυρία Πετήρ και βλέπουμε. Πρόεδρε, καταρχάς μπερδεύτηκα το Ποιος ζήτησε αυτή την έκθεση. Η Επιτροπή Γεωργίας, ποιος από εμά το ζήτησε. Είναι εδώ εκείνος που ζήτησε αυτή την μελέτη, να ακούσει. Ίσως τελικά πρέπει να βγάλουμε άκρη με αυτό. Ίσως προήλθε από την αριστερά του σώματος. Θεώρησε ότι υπήρχε κάποια συνωμοσία με πολύ κακές σατανικές εταιρείε που παίρνουν το φαΐ από το στόμα του καταναλωτού και τα κέρδη από τα χέρια των αγροτών. Αυτό όμως που είδα είναι ότι το κόστος να διατεθεί φυτοποσταστικό υλικό στην αγορά από 152 εκατομμύρια δολάρια πήγε στα 256 εκατομμύρια δολάρια. Τεράστια αύξηση. Και μόνο οι πιο δυνατοί μπορούν να αντέξουν αυτό το κόστος. Αν υπήρξε κάποια συγκέντρωση εταιριών λοιπά, μεγάλων στον τομέα αυτό, να η απάντησή σας. Μόνο οι πιο δυνατοί, οι πιο μεγάλοι μπορούν να το κάνουν. Και ποιος θα έκανε πολύ δαπανηρό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέβασε τις τιμές τόσο. Η η μερίσια διάταξη ε, εξετάζεται και καθορίζεται από τους συντονιστές. Ίσως ήσταν απόν στη συνεδρίαση που κανονίσαμε την ημερησία διάταξη. Αλλά ρωτήσατε ποιος ζήτησε την ε, εκπόνηση αυτής της μελέτης και σε ποιον πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Καλώς. Τα συγχαρητήριά σας ε, στον εμπνευστή αυτής της μελέτης θα τα μεταφέρω στους συντονιστές. Εγώ πιστεύω πάντως ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Κύριε Πετήρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι η τρίτη τέταρτη μελέτη που έχουμε ακούσει το τελευταίο 1,5 χρόνο από τότε που είμαι και εγώ ευρωβουλευτής και ούτε σε μία από αυτές τις μελέτες δεν αναφέρεται η Κροατία που είναι πια πλήρες μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και δύο χρόνια. Γιατί λοιπόν δεν λαμβάνετε υπόψη τα στοιχεία σας και την Κροατία θα ήθελα να ζητήσετε από τις υπηρεσίες, στις ε, μελλοντικές αναλύσεις και μελέτες, να λαμβάνετε υπόψη και στοιχεία από την Κροατία που είναι πλέον πλήρες μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε απόλυτο δίκιο κυρία Πέτυρ. Φυσικά, όλες οι χώρες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όλες οι χώρες να δίνουν τα στοιχεία τους σε τέτοιες μελέτες. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαβάσατε με μεγάλη ταχύτητα τους αριθμούς, άλλωστε οι βουλευτές προτιμούν να έχουν συμπυκνωμένα τα συμπεράσματα εν τέλει. Τέλος πάντων το να μεγαλώνει ε, μια επιχείρηση, ένας όμιλος επιχείρησεων δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό από την άλλη μεριά μπορεί να οδηγήσει σε δεσπόζουσα θέση στην αγορά εφόσον προκύπτουν μονοπόλια. Στους τομείς με τους οποίους περάσατε με τέτοια μεγάλη ταχύτητα εντοπίσατε κάποιες ανησυχητικές τάσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μονοπόλια, κάτι το οποίο δεν είναι καλό βέβαια για την οικονομία. Διότι οι μονοπόλια σημαίνουν υψηλότερα κέρδη για τις επιχειρήσεις, μεγαλύτερες υψηλότερες τιμές δηλαδή για την γεωργία. Κύριε Βουλευτά, ε, η μελέτη είναι πολύ πιο εκτεταμένη και έχουμε την πλήρη μελέτη στη διάθεσή μας. Θα έχετε όλο το χρόνο στις διακοπές να εντρυφήσετε σε ολόκληρη τη μελέτη. Νίκολσον. Ε, ο κύριος Γιάρμπου είναι σαν και εμένα, τα αφήνει όλα για τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Μπορεί να είμαστε ολίγοι, αλλά είμαστε πολύ μεγαλόκαρδοι. Και θέλουμε να φτάσουμε στο τέρμα της εργασίας μας. Εδώ και κάνα δύο χρόνια όταν έκανα ομιλίες αναφερόμαστε στα τρία F στα αγγλικά. Ζωοτροφές, κάψιμα και λιπάσματα. Και λέγανε ότι ήταν υψηλές οι τιμές το και γι' αυτό ήταν υψηλές οι τιμές των προϊόντων οι τιμές των καψίμων επηρέασαν τα λιπάσματα. αυξήθηκε η τιμή των λιπασμάτων, μας είπαν τότε λόγω των καυσίμων του βαρελιού του ε, πετρελαίου τελικά δεν επανήλθε η τιμή του πετρελαίου παρά που ε, δεν μειώθηκε η τιμή του λιπάσματος παρόλο που μειώθηκε η τιμή του πετρελαίου. Κάπως κάποιος πρέπει να εκτεθεί γιατί βγάλει πολύ μεγάλα κέρδη. Διότι αν έβγαλαν τα κέρδη που έβγαζαν πριν ανέβει όταν ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου και τώρα έχει κατέβει η τιμή αλλά δεν έχουν μειωθεί οι τιμές των προϊόντων, κάποιος βγάζει μεγάλα κέρδη. Δεν θέλω να κάνω αστεία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η αντιμετώπιση, ε, το κόστος της ε, παραγωγής προϊόντων από τους γεωργούς σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει άλλος κανείς το λόγο. Φυσικά, ε, οι τιμές αυτές ε, επηρεάζουν το γεωργικό εισόδημα. Γιατί πολλές φορές ε, η τιμή ενός λίτρου γάλακτος ε, συνδυάζεται με την τιμή που είχε ένα λίτρο λαδιού ή νερού. Είναι όλοι ε, αυτοί οι συντελεστές σημαντικοί στη διαμόρφωση των γεωργικών τιμών. Ακούσατε τις ερωτήσεις, έχετε το λόγο παρακαλώ για να απαντήσετε. Ναι. Γρήγορες απαντήσεις προς την Κροατία δεν είχαμε τα στοιχεία από το δίκτυο, στο δίκτυό μας διαθέσιμο από την Κροατία. Πρόσφατα έγινε μέσα Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κροατία. Την επόμενη φορά θα το κάνουμε. Δεν είναι ότι δεν είχαμε παρατηρήσει ότι τα μέσα Ευρωπαϊκή Ένωση η Κροατία ήταν δύσκολο να συμπεριλάβουμε τότε τα στοιχεία που αφορούσαν την Κροατία. Το γενικό ερώτημα όσον αφορά αυτό που έθεσε ο συνάδελφος του Ηνωμένου Βασίλειο. Πράγματι, βλέποντας τα ποσοστά συγκεντρώσεως βάσει της μελέτης μας, δεν βλέπουμε τομείς όπου θα έπρεπε να ανησυχούμε υπερβολικά για συγκεντρώσεις. Αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η καινοτομία σε κάποιους τομείς όπως των σπόρων και στα, στον τομέα της πιστοπροστασίας μειώθηκε βλέποντας τα διάφορα στοιχεία όσον αφορά την ευρεσιτεχνία. Δηλαδή για να εγκριθούν τα προϊόντα για διάθεση στην αγορά απαιτείται πολύ μεγάλη, μεγάλο τίμημα, το κόστος παίζει μεγάλο ρόλο, έχουμε ρυθμιστικό εμπόδιο λοιπόν. Είναι ένας φραγμός που στηρίζει τη συγκέντρωση στους τομείς, διότι οι μικρότερες εταιρείες δεν μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά εύκολα. Αυτό ισχύει μόνο για εταιρείες που παράγουν χημικά προϊόντα και προϊόντα για τον έλεγχο των φυτών και επίσης και για εταιρείες που παράγουν βιολικά τέτοια μέσα. Υπάρχει μεγάλο κόστος για την έγκριση των προϊόντων. Οπότε η είσοδος τους στην αγορά περιορίζεται λόγω αυτών των εμποδίων. Αν υπάρχουν τάσεις που μας ανησυχούν, συμπεράναμε στη μελέτη μας ότι όσον αφορά τις παρατηρούμενες συγκεντρώσεις δεν υπάρχει ουσιαστική τάση που να μας ανησυχεί. Υπάρχουν κάποιοι μικροί τομείς της αγοράς όπου τα ποσοστά συγκέντρωσης είναι υψηλότερα από τις άλλους τομείς. Αυτό εξηγείται διότι είναι αγορές πολύ περιορισμένες και αν πούμε ότι εκεί χρειάζεται με ανταγωνισμός δεν υπάρχει περιθώριο τόσο μικρές οι αγορές και εκεί δρούν δύο-τρεις εταιρείες ε, και επενδύουν οπότε δεν θα ήταν χρήσιμο διότι η κοινωνική ευημερία θα μειωνόταν όσον αφορά τα τρία F που αναφέρατε και τα μονοπόλια στις αγορές των λοιπασμάτων ή τις αλλαγές όσον αφορά τις τιμές των ε, λοιπασμάτων σχετίζονται οι τιμέ των λιπασμάτων πολύ με τι αλλαγέ τη τιμή του πετρελαίου. Αυτό είναι πασίγνωστο. Όταν μειώθηκαν οι τιμέ του πετρελαίου, γιατί δεν είδαμε μια μείωση στην τιμή των λιπασμάτων, όπω αναφέρθηκε. Τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μα, παρατηρήσαμε μια μείωση στην τιμή των λιπασμάτων. Μπορεί να συζητήσει κανεί κατά πόσο η τιμή τη τιμή των λιπασμάτων ήταν τόσο μεγάλη όσο και η μείωση τη τιμή του πετρελαίου. Βλέποντας τα αυτά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν έγινε η μείωση στο ίδιο ποσοστό. Ξέρουμε όμως πάντα ότι υπάρχει κάποια υστέρηση όσον αφορά την ανταπόκριση κάποιων βιομηχανιών. Αν κάποιος έβγαλε υπερβολικά κέρδη στον τομέα, δεν μπορούμε να κρίνουμε συναρτήσει των διαθεσίμων στοιχείων. Τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η συγκέντρωση στον τομέα των λοιπασμάτων δεν είναι τόσο υψηλή οι εταιρείε λοιπασμάτων, εάν υπήρχε μεγαλύτερη συγκέντρωση θα είχαν δυνατότητα σχεδόν μονοπωλιακή στον καθορισμό των τιμών. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, μπορώ με τα χαρά να απαντήσω μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν έχετε άλλες απορίες και με τα χαρά να σας απαντήσω. Σας ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη. Όντως είναι περίπλοκη η πραγματικότητα και αυτό το διαπιστώνουμε και στις συζητήσεις που έχουμε με τους γεωργούς. Όταν μιλούμε για τις ενισχύσει και για τα εισοδήματά τους. Πολύ χρήσιμη πάντως αυτή η μελέτη. Καταφέραμε και διεκπαιρεώσαμε την απογευματινή μας ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονές μας για την παρουσίαση. Και φυσικά σας συνιστώ την ενδελεχή ανάγνωση αυτής της μελέτης στον ελεύθερο σας χρόνο. Και μην ξεχνάτε και τη χριστουγεννιάτικη δεξίωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Γεωργών που όπως ε, σας είπα θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρα συνεδρίες 6.30 στο ίδιο κτίριο, στο εστιατόριο ο κύριος Φλάναγκαν όταν ε, έχετε παρουσίαση με powerpoint ή με διαφάνειες θα φροντίζετε να μοιράζετε τις διαφάνειες εκ των προτέρων στους ευρωβουλευτές. Γιατί κάνω ό,τι μπορώ για να κοιτάξω τη μεγάλη οθόνη, αλλά δεν έχω και βιονικά μάτια για να τα διακρίνω όλα. Οπότε, αν δεν μας στέλνετε τις, ε, τα, σχετικά, ε, τα σχετικά έγγραφα, τουλάχιστον να τα φροντίζουμε εμείς να τα στέλνουμε γιατί έχουμε τόση πολύ τεκμήριωση και της COP21, ε, θα, ε, αν το συγκεντρώνουμε όλα αυτά σε έγγραφα, θα είχαμε ε, έγγραφα μέχρι τον πύργο του Άιφελ ψηλά. Να μην ξοδεύουμε χαρτί. Παρακαλώ θα, το, θα ενημερώσω τη γραμματεία και θα το αναλάβει. Επαναλαμβάνω, μην ξεχνάτε την πρόσκληση για τη χριστουγεννιάτικη δεξίωση των νεαρών γεωργών στο κτίριο που βρισκόμαστε στο εστιατόριο. Καλώς βράδυ.